La séance est ouverte. Euh, Αρχίζει η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Ησυχία παρακαλώ. Όσοι είναι εκεί πίσω όρθιοι στα πηγαδάκια, παρακαλώ ή καθίστε ή αποχωρήστε. Έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Έχω κάποιες ανακοινώσεις στο σημείο 2 όσον αφορά τις γλώσσες. Οι γλώσσες είναι οι συνήθεις που χρησιμοποιεί η Επιτροπή μας ανάλογα με τις ανάγκες των μελών. Τα έγγραφα συνεδρίασης έχουν ε, διανεμηθεί μέσω διαδικτύου βάσει της πολιτικής μας που είναι να μην έχουμε καθόλου ε, έγγραφα σε χαρτί. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει αναμετάδοση μέσω διαδικτύου και μας ακούνε δηλαδή μέσω διαδικτύου. Επίσης θέλω να σας πω ότι από την 21η Μαρτίου τα έγγραφα της ομάδας κώδικας δεντολογίας είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα συμβουλευτείτε σε μια αίθουσα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίπλα στα γραφεία του προσωπικού της Επιτροπής Τάξα στην πλατεία Ντεμέους. Εγώ ίδιος πήγα εκεί ήδη από τις πρώτες μέρες και πολλοί από εσά έχουν επίσης πάει. Σας υπενθυμίζω τα ωράρια. Πότε μπορείτε να συμβουλευτείτε τα εγγραφέ εκεί είναι Δευτέρα με Πέμπτη 9 με 12.30 το πρωί και 9.30 με 5.30 το απόγευμα και τις Παρασκευές 9 με 12.30. Βέβαια πρέπει προηγουμένως να έρθετε σε επαφή με την γραμματεία έγκαιρα για να... Μέχρι τέσσερις μπορούν συγχρόνως να συμβουλευτούν έγγραφα εκεί ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι αποφάσισαν οι συντονιστές. Κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε με τους συντονιστές των ομάδων για να κάνουμε τον πρώτο απολογισμό. Τώρα, τα καλά νέα όσον αφορά την προετοιμασία της διακοινοβουλευτικής μας συνάντησης στις 18 Απριλίου. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, καλέσαμε εκπροσώπους των ορμοδίων επιτροπών των 28 κοινοβουλίων των χωρών μελών και έχουμε ήδη 35 βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν εγγραφεί για αυτή τη συνάντηση από 20 περίπου Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο σημείο 3, θέλω να αναφερθώ λίγο στο Panama Papers, αυτή την υπόθεση στην οποία εδώ και δύο μέρες αναφέρεται συνέχεια ο τύπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει αν θέλει να αντιδράσει στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, ότι είναι μια υπόθεση που θα έχει συνέπειες για όλες τις αρχές οι οποίες καλούνται να λάβουν φορολογικές αποφάσεις και θα πρέπει να κάνουν έρευνες, ελέγχους και προτάσεις. Μεταξύ άλλων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δικιά μας Επιτροπή Τάξη 2, συνεπώς. Μίλασα λίγο με τον Γέπε Κοφούτ, που είναι ο εισηγητή μας. Ο Μάικλ Τάουερ, ο οποίος ε, είναι συνεισηγητής, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί είναι στην κηδεία του Κίτο Φαστεβέλε, στη Γερμανία. μεταφέρουμε στην οικογένεια του αποθανόντος τα συλληπιτήριά μας. Διαπιστώσαμε πάντως με τον Γέπε ότι όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων, για να μην πω εκατομμύρια, τα οποία θα αποκαλυφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, θα πρέπει με τους συντονιστές να καθίσουμε και να συζητήσουμε ε, τα συμπεράσματα στα οποία πρέπει να καταλήξουμε όσον αφορά τις δικές μας τις έρευνες, το δικό μας το έργο και να λάβουμε υπόψη μας τις αποκαλύψεις αυτές είτε στα πλαίσια της Επιτροπής μας τάξη 2 είτε σε ένα άλλο πλαίσιο. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Να γνωρίζετε πάντως ότι το Προεδρείο του ΤΑΞ 2 και οι συγκητές το καταλαβαίνουν αυτό. Έχουμε προβλέψει να συνεδριάσουμε στις 18 Απριλίου οι συντονιστές μετά την διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Νομίζω ότι είναι καλή στιγμή εκείνη, γιατί τότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Αν μη τι άλλο θα ξέρουμε ποιες είναι οι πληροφορίες αυτές που θα έχουν αποκαλυφθεί. Και έτσι σε επίπεδο συντονιστών, αλλά και Επιτροπής ΤΑΞ 2, να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Τώρα λοιπόν περνάω στο σημείο 3 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Φεστάγερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαργαρέτ Φεστάγερ που είναι στη διάθεσή μας και πάλι να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας. Θέλω να τη συγχαρώ για το θάρρος της στη μάχη αυτή που δίνει σε ένα τομέα πολύ σημαντικό αλλά συγχρόνως και πολιτικά και νομικά πολύ λεπτό. Είναι ο έλεγχος των κρατικών ε, επιχορηγήσεων μέσω της φορολογίας. Η δράση της, δίχως άλλο, συνάδει απόλυτα με τις προτάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Επιτρόπου Μοσχοβησή. Είναι οι προτάσεις που έχει θέσει η Επιτροπή επιτάπητος στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ και λαμβάνονται υπόψη και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συστάσεις που έχουμε εγκρίνει στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και για την έκθεση τη επιτροπή ΤΑΞ 1, αλλά και γενικότερα με τις εκθέσει και τα ψηφίσματα που έχουμε εγκρίνει. Θα μας παρουσιάσετε λοιπόν το πρόγραμμά σας για το έργο σας τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουμε την παράδοση που έχουμε στην Επιτροπή αυτή. Δηλαδή 10 λεπτά θα μας παρουσιάσετε εσείς ε, τη θέση σας, τα δρόμενά σας και μετά θα πάρουν το λόγο εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν που με προσκαλέσατε εδώ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ε, Είμαι πολύ ικανοποιημένη που αποφασίσατε να συνεχίσετε την ε, δουλειά αυτή. Νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό για την συνέχεια της ε, πρώτης επιτροπής για την φορολογία και για να εμβαθύνετε από αυτό απαιτείται. Εκτιμώ τη δουλειά που έχετε κάνει. Νομίζω πως παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής γενικώς αλλά και βεβαίως το να διατηρηθεί μια δυναμική για να επέλθει η αλλαγή. Ο στόχος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής σας Επιτροπής νομίζω πως ε, είναι σχεδόν ταυτόσιμος. Εμείς στην Κομισιόν θέλουμε μια δίκαιη εταιρική φορολογία και βεβαίως αυτό βασίζεται κυρίως στην αρχή του να έπανα συσταθεί η σύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας με την ε, φορολογία. Και βέβαια όταν λέμε για τα πράγματα τόσο απλά αρχίζουν μετά τα περίπλοκα. Γιατί πώς γίνεται κάτι τέτοιο είναι το ερώτημα. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα βρούμε και εμείς ε, και οι ειδικοί γιατί νομίζω πως έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο από τον Σεπτέμβριο πέρσι τον Ιανουάριο, λοιπόν, προτείναμε να κλείσουν κάποια σημαντικά παραθυράκια που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να μην πληρώνουν φόρους. Επίσης, προτείναμε οι πολυεθνικές να αποκαλύπτουν τα φορολογικά τους στοιχεία στις ε, φορολογικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν σημείο της ε, σημασίας ε, της πρότασης αυτής ότι υπάρχει ήδη μία πολιτική συμφωνία υπό την αίρεση βεβαίως του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τις ε, μελέτες επιπτώσεων για να αυξηθεί η διαφάνεια στην εταιρική φορολογία. Επίσης έχουμε προχωρήσει αρκετά όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού όσον αφορά τους ε, κανόνες ε, κρατικών ενισχύσεων. Ανακαλύψαμε πέρσι πως η Fiat και η Starbucks είχαν αδικαιολόγητα φορολογικά πλεονεκτήματα. Το Δεκέμβριο ανοίξαμε μια έρευνα για το εάν το Λουξεμβούργο έκανε μια ρύθμιση με τη McDonald's που δεν ήταν διαθέσιμη σε άλλες εταιρείε. Τον Δέη Ιανουάριο βρήκαμε πως το σχετικό σύστημα του Βελγίου ήταν παράνομο και ζητήσαμε μια ανάκτηση 700 εκατομμυρίων ευρώ από 30 εταιρείες. Στις ε, τελευταίες περιπτώσεις δε είχε ξεκινήσει η διαδικασία της ανάκτησης, για την Fiat έχει ολοκληρωθεί κιόλα. Το Λουξεμβούργο έχει ανακτήσει το σύνολο των ασύμβατων ενισχύσεων από την Fiat. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι γνωστές, τα έχουμε ξαναπεί. Οπότε σήμερα θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά ελπίζω να είναι εξίσου σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια εξετάσαμε πάνω από χίλιες τέτοιες μεμονωμένες φορολογικές αποφάσεις. 600 από αυτές ήταν από τα LuxLeaks. Οι υπόλοιπες προέκυψαν από τις δικές μας έρευνες που ξεκίνησαν το 2013 και επεκτάθηκαν ε, στο τέλος του 2014 σε μια συστηματική εξέταση των αποφάσεων αυτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν σταδιακά. Πρώτα απ' όλα ζητήσαμε από όλα τα κράτη-μέλη έναν κατάλογο όλων των αποφάσεων που είχαν λάβει υψηρά ετών και με τη βάση αυτή Ζητήσαμε τις μεμονωμένες αποφάσεις από εταιρείε που επιλέξαμε από τον κατάλογο που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα βεβαίως ήμασταν πολύ προσεκτικοί με τις μεγάλες εταιρείε και τις εταιρείε που είχαν τις πιθανότητες να είναι οι λεγόμενοι εθνικοί πρωταθλητές. Δηλαδή αν ε, θα έκανε κάποιος μία χάρη θα ήταν στις μεγάλες εθνικές εταιρείε. Κάναμε την ε, δουλειά μόνοι μας ε, με μια ομάδα από ειδικού στα νομικά και την φορολογία από την Κομισιόν και τις Εθνικές ε, Φορολογικές Διοικήσεις. Εκεί όπου δεν ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, ζητήσαμε διευκρινήσεις από τα κράτη-μέλη. Τώρα γνωρίζουμε πως όλα τα κράτη-μέλη πλην πέντε εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή πλην της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Κροατίας, της Λετωνίας και της Σλοβενίας. Και δεν είναι με αλφαβητική ε, σειρά. Δεν χρησιμοποιούν λοιπόν καθόλου φορολογικές συμφωνίες αυτές οι χώρες. Τα 23 κρατημέλη που χρησιμοποιούν φορολογικές συμφωνίες, κάποια κάνουν μόνο κάποιες λίγες συμφωνίες το χρόνο, αλλά κάνουν χιλιάδες. Και τώρα έχουμε πολλές ενδείξεις για το πώς ε, τις χρησιμοποιούν αυτές. Τα καλά νέα είναι πως οι περισσότερες από αυτές τις ε, συμφωνίες δεν αφορούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Παραδείγματο χάρη, στο LuxLeaks πρόκειται κυρίως για αποφάσεις ε, επιβεβαιωτικές όπως λέμε. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ απλές, δεν περιέχουν καθόλου υπολογισμό των κερδών. Ρωτάνε μία ερώτηση και τους απαντάνε με ένα ναι ή με ένα όχι. Και άρα έτσι δεν ε, τίθεται ζήτημα κρατικών ε, ενισχύσεων γιατί δεν κάνουν και πολλά πράγματα οι φορολογικές αρχές, αλλά ε, αυτό ίσως δεν ισχύει για όλες τις επιβεβαιωτικές τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό ακριβώς εξετάζουμε την περίπτωση των McDonald's. Πολλές αποφάσεις ακολουθούν την ε, πολύ βασική αρχή ότι θα πρέπει τα κέρδη να φορολογούνται εκεί όπου δημιουργούνται. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο, ειδικά όταν έχουμε προχωρημένες πρακτικές τιμολόγησης με transfer pricing ε, μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου σε διαφορετικές χώρες ή μεταξύ εταιριών που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Γύρω στις 200 ε, αποφάσεις από αυτές που έχουμε ζητήσει έχουν τέτοια μορφή. Το transfer pricing δεν είναι προβληματικό εάν ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ανταποκρίνεται δηλαδή σε τιμές οι οποίες φαίνονται σε παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ εταιριών που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οπότε η πρακτική καθ' αυτή δεν είναι προβληματική, αρκεί να γίνεται μια πραγματική προσπάθεια να αντιστοιχούν οι τιμές με την οικονομική πραγματικότητα. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα λοιπόν με τις ε, βέλτιστες πρακτικές μπορούν τα κράτη-μέλη να είναι σίγουρα πως οι συμφωνίες αυτές αντικατοπτρίζουν όντως την οικονομική πραγματικότητα. Και η έρευνά μας έδειξε ότι πολλές τέτοιες αποφάσεις δεν εγείρουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Όμως, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, βρήκαμε περιπτώσεις πολύ πιο ανησυχητικές, όπου έχουμε τέτοιες αποφάσεις που χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να ευνοήσει συγκεκριμένες εταιρείες ή ήδη εταιρεών. Οι υπηρεσίε μου θα εξετάσουν αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς τους επόμενους μήνες, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια ιδέα των προβλημάτων που έχουμε. Πρώτα απ' όλα, κάποιες ε, συμφωνίες ε, γύρω στις 100 ε, κοιτούν μόνο την μία πλευρά της ε, συναλλαγής και αποφασίζουν μετά για το κατάλληλο κέρδος ε, με βάση μία μόνο εταιρεία του ομιλός αφορά το κέρδος το οποίο απομένει μπορεί να φορολογείται κάπου αλλού ή να μην φορολογείται καθόλου. Και έτσι δημιουργείται η δυνατότητα να υπάρχουν παραθυράκια. Δεύτερον, έχουμε την ε, ανησυχία για την χρηματοδότηση για τις ε, εταιρείε ε, χαρτοφυλακίου που μόνος τους ρόλος είναι να δανείζονται χρήματα από μία εταιρεία του ομίλου και να τα δανείζουν σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί η φορολογητέα ύλη. Οπότε, μέχρι στιγμής είχαμε εξετάσει το transfer pricing, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών ε, φορολογικές αποφάσεις. Όπως είπα, κάποιες αποφάσεις απλά επιβεβαιώνουν το εάν ένας κανόνας ισχύει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίω ε, πρόκειται έτσι για μια αποτύπωση μιας στιγμής. Ε, πιθανών ανησυχιών και των, διατάκ, των με διαστάσεων που προανέφερα, δεν μπορεί να προδικάσει πιθανές νέες προβληματικές περιπτώσεις. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεύτερο, σήμερα, ε, είναι το δικό σας το αίτημα για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα προλάβουμε και θα αποτρέψουμε το να γίνει η εφαρμογή του φορολογικού δικαίου ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρώτα απ' όλα, όταν δημοσιεύονται οι αποφάσεις μας, ε, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις ε, εταιρείες, αλλά κάτι άλλο τον Ιούνιο θα συναντήσουμε τους ειδικού από τα κράτη-μέλη στο Φόρουμ Φορολογίας Υψηλού Επιπέδου για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες στην πράξη. Και για να στηρίξουμε αυτή την συζήτηση θα δημοσιεύσουμε ένα έγγραφο εργασίας που θα περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες για αυτά τα οποία έχουμε μάθει από τις χίλιες ε, τέτοιες ε, συμφωνίες. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα το καινούριο. Δεν πρόκειται για καμιά αποκάλυψη λοιπόν. Πρόκειται για παλαιού τύπου ευρωπαϊκή νομολογία. Το δικαστήριο έχει ξεκαθαρίσει από δεκαετία του 1970 ότι οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων ισχύουν για τις φοροαπαλλαγές, όπως ακριβώς και οι άμεσες κρατικές ενισχύσεις. Προφανώς. Είτε σου δίνουν λεφτά, είτε πληρώνεις λιγότερους φόρους, το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Βεβαίως, ε, η στρέβλωση είναι επίσης η ίδια, εάν είναι επιδότηση σε μετρητά ή λιγότερη φόρη. Υπήρχε επίσης και η απόφαση του 2006 για το Βέλγιο, όπου επιβεβαιώθηκε το ότι η αρχή την οποία προανέφερα για την σύγκριση με ανεξάρτητες συναλλαγές είναι αυτή η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αν δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα πλέον εκτήματα δηλαδή, για συγκεκριμένες εταιρείες, π.χ. εάν αυτή η εξαίρεση είναι διαθέσιμη σε όλες τις εταιρείες, τότε δεν τίθεται ζήτημα κρατικής ενίσχυσης. Οπότε, όσο σωστά και αν εφαρμόσουμε τους κανόνες, πρέπει να βελτιώσουμε και το φορολογικό δίκαιο στο εθνικό και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν γίνεται εν κενό. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί για συνεργασία μαζί σας με το Συμβούλιο και βεβαίω με τους εταίρους μας του ΟΣΑ και των G20. Γι' αυτό θεωρώ πως η Επιτροπή ε, τάξε 2 τώρα θα περάσει στην επόμενη φάση του έργου της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Merci beaucoup, Madame le Commissaire. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους διάφορους ομιλητές για πεντάλεπτες ε, ερωταπαντήσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Κόφοντ, που είναι συνεισηγητής και εκπρόσωπος της ομάδας των σοσιαλιστών. Για Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Επίτροπε θα έπρεπε να σας απευθύνω το λόγο στα Δανέδικα, αλλά θα μιλήσω αγγλικά. Καταρχάς θα ήθελα να πω και εξ ονόματος των συναδέλφων, όπως και ο Πρόεδρος, να εκφράσω την μεγάλη μας εκτίμηση για την εργασία που κάνετε στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ανταγωνισμού με αυτές τις υποθέσεις, ε, προσπαθώντας να εξασφαλίσετε το δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς επίσης και να εντοπίσετε τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις και τα tax rulings. Αυτό που είδαμε σήμερα και χτες βέβαια με τα έγγραφα του Παναμά και όλο το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από αυτό δείχνει ότι αν κανείς φωτίσει όλα αυτά τα πράγματα αυτό που διαπιστώνει είναι ότι υπάρχει σχεδιασμός φορολογικός, επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και φοροαποφυγή ε, και γι' αυτό και η δική σας εργασία είναι τόσο σημαντική. όλες οι υποθέσεις που έχει αναφέρει η Κομισιόν, όπως η Starbucks στην Ολλανδία, η Fiat ε, στη Λουξεμβούργο. Η ερώτησή μου είναι πώς επιλέγει η Κομισιόν ποιες υποθέσεις θα αναλύσει περισσότερο και ποια μέτρα λαμβάνει ώστε να εξασφαλίσει ότι θα επιβληθεί καταλήλως ο νόμος για όλους. Αναφερθήκατε στις ε, κατευθύνες γραμμές, είναι πολύ σημαντικό και έπειτα αναφέρετε στην αρχή της, ε, την ε, δημόσια συζήτηση για τις αναχώρα εκθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό για όλες τις χώρες εντός και εκτός Ένωσης, διότι αν δεν έχουμε σωστή συζήτηση για όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς η ε, συμπολίτε μα, κάποιοι συμπολίτε μα προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Ευχαριστώ. Η κυρία Επίτροπο. Για το θέμα του ποιε υποθέσει ανοίγουμε και εξετάζουμε. Καταρχάς, μάλλον να ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σας λόγια. Ορισμένα αυτά θα τα απευθύνονται κανονικά στον προηγούμενο επίτροπο, στην επόμενη, προηγούμενη επιτροπή, γιατί πολλές από αυτές τις υποθέσεις ε, τις άνοιξε ο συνάδελφος Αλμούνια. Και τα συγχαρητήρια αξίζουν και στα κοινοβούλια που κάνουν πολλή δουλειά, ε, συγκαλούν δημόσιες ακροάσεις ώστε να ε, χυθεί φως σε όλες αυτές τις φορολογικές ειδικέ ρυθμίσεις. Γιατί αυτοί αποτέλεσαν την έμπνευση ώστε να ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις. Ε, ξεκίνησαν από πρωτοβουλίες βουλευτών όλα αυτά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν δεν είναι κάτι που μια εταιρεία ας πούμε, διαμαρτύρεται κατά μια άλλη εταιρεία, αλλά κανεί δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Παρότι αυτό μα προκαλεί απορία. Να πει δηλαδή ότι κοιτάξτε, αυτοί εκεί ε, αποφελούνται από ένα ειδικό φορολογικό καθεστώ. Ανοίγουμε λοιπόν τις υποθέσεις ε, όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για ανησυχία. Προφανώς μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις υποθέσεις, αλλά μόνο αυτές που πιστεύουμε ότι υπάρχει βάσιμη ε, λόγος για ανησυχία. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Γιατί βεβαίως μπορεί να φανταστείτε ότι η φαιά είναι ε, μεγάλη. Υπάρχουν εταιρείε που δεν αμφισβητούνται βέβαια και κράτη που δεν αμφισβητούνται, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη φαιά ε, ζώνη ε, όπου προσπαθούμε να βρούμε τις πιο ανησυχητικέ ε, περιπτώσεις και υποθέσεις. Και βεβαίως προσπαθούμε να καλύψουμε και διάφορους τρόπους παροχής αυτών των επιλεκτικών πλέον εκτιμάτων που σας είπα. Έχουμε κάνει διάφορες υποθέσεις μεταφοράς ε, δήλωση των κερδών ή περιπτώσεις όπου έχουμε ε, συγκεκριμένα στοιχεία για την αναχώρα, τις αναχώρα εκθέσεις. Θα το συζητήσουμε ε, σύντομα στην Κομισιόν. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Βεβαίως, από τη μία πλευρά θα πρέπει να σεβαστούμε τη δικαιοδοσία μας. Και βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πνίξουμε γραφειοκρατικά τις εταιρείε. Ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες και στο σωστό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να γνωρίζει το κοινό, να γνωρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως ε, να αλλάξει όλη η νοοτροπία σε σχέση με τη φορολογία. Ευχαριστώ πολύ. Brian Ace. Brian. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε, στην Επιτροπή ΤΑΞ 2 και σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που κάνετε και για την υπευθυνότητα που έχετε δείξει από τότε που οριστήκατε σε αυτή τη θέση. Εξετάσατε διάφορες υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί φορολογικές αποφάσεις. Για την υπόθεση της Apple τι θα γίνει. Ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν, αλλά ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα έχουμε απόφαση. Μας δώσατε και μια σημαντική πληροφορία. Είπατε ότι για τις ρυθμίσεις αυτές 200 έχουν να κάνουν με θέματα ε, μεταβίβασης ε, τιμολόγησης. Πόσες χώρες ερευνώνται για αυτό το θέμα και πόσες είναι από τις 200 αυτές που αναφέρατε. Τρίτον, για το θέμα των εγγράφων ε, από τον Παναμά. Κύριε Επίτροπε, σε αυτό το στάδιο που είναι βέβαια πολύ πρόωρο, γνωρίζετε μήπως καθόλου αυτές οι νέες πληροφορίες πώς συνδυάζονται με κάποιες από τις έρευνες που ήδη έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ίσως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει τέτοια διασταύρωση. Και πώς θα ενημερωθούμε εμείς. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη μετά από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις να αρχίσει νέες διαδικασίες, νέες έρευνες κατά συγκεκριμένων εταιριών που κατονομάζονται στις πληροφορίες αυτές που τώρα βγαίνουν. Και τέλος, κύριε Επίτροπε, έχουμε ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε την νομοποίηση παράνομου χρήματος και άλλες οδηγίες. Όλα αυτά πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάποια διάκριση ανάμεσα στις τρίτες χώρες και την διαφθορά αυτή καθεαυτή που φαίνεται μετά από τις αποκαλύψεις Παναμά. Ευχαριστούμε. Η Επίτροπος να απαντήσει. Ευχαριστώ. Για την Apple, όπως και για οποιαδήποτε άλλη, ισχύει το ίδιο. Ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η ποιότητα της δουλειάς μας. Οπότε ακολουθούμε τις διαδικασίες. Άμα έχουμε νέες πληροφορίες, τίθενται νέα ζητήματα και αυτά τα νέα ζητήματα πρέπει να πάνε πίσω στις χώρες μέλη και μερικές φορές και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προγνωστικά, να πούμε δηλαδή πότε θα είμαστε έτοιμοι για απόφαση. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Apple. Χρειάστηκε να ζητήσουμε νέες πληροφορίες, κάτι το οποίο ανέβαλε βέβαια την ολοκλήρωση του ζητήματος και την κατάληξη. Τώρα όσον αφορά το transfer pricing. Από τα νούμερα δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα για το πόσες θα είναι οι προβληματικές περιπτώσεις, γιατί μερικές φορές αυτό το transfer pricing γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες. Δηλαδή αντικατοπτρίζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα, υπάρχουν τα σωστά έγγραφα. Αυτό όμως το διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες μέλη. Και για αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλουμε να μην προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό και σήμερα ζητήσαμε να υπάρξει αυτή η συνάντηση υψηλού επίπεδου, ώστε ακόμα και αν είναι πρόημο να δώσει κανείς κατευθυντήριες γραμμές, αν μη τι άλλο να μπορέσουμε τις χώρες μέλη να συζητήσουμε σε βάθος ώστε να μην προκύπτουν νέες τέτοιες περιπτώσεις. Μόνο τις καλές πρακτικές να τις ε, ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι χώρες μέλη. Αυτό ναι. Για τα Panama Papers, για τα έγγραφα αυτά που προέκυψαν από τον Παναμά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Από ό,τι λίγο είδα, έχει να κάνει με επιχειρήσεις και από άτομα τα οποία οργανώνονται ε, με επιχειρήσεις offshore δεν φαίνεται να τίθεται θέμα κρατικών επιχορηγήσεων. Μπορεί να τίθεται θέματα φορολογικά γενικά, ναι. Ένα από τα παράδοξα είναι ότι μέρος αυτών των δραστηριοτήτων είναι νόμιμες. Μπορεί να μην είναι σωστές, αλλά είναι νόμιμες. Και αυτό είναι ζήτημα για τον νομοθέτη. Να δει τι θέλουμε τελικά να κάνουμε. Η συζήτηση αυτή βρίσκεται στα πρώτα μόλι στάδια. Αν γίνει συζήτηση θα ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Προς το παρόν δεν ξέρω κατά πόσο αποκαλύψεις αυτές θα αλλάξουν τις έρευνες που ήδη είναι σε εξέλιξη ή θα μας οδηγήσουν να αρχίσουμε και νέες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Βέρνερ Λάγκεν. Για τα Panama Papers σίγουρα για τις αποκαλύψεις αυτές. Θα μας δώσετε ένα αντίγραφο αυτού που έχετε στα χέρια σας, έτσι. Πολλά τεραμπάιτ. Λέει ο κύριος Λάγκη, εκτός μικροφώνου, όμως δεν ακούμε καλά. Τι Μπορζάνη, εκ μέρους των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις οι οποίες όμως δεν συνδέονται μεταξύ τους. Υπό το φως του σκανδάλου του Παναμά και ίσως και κάποιων προηγουμένων υποθέσεων, πιστεύω ότι ο αγώνας μας κατά των φορολογικών παραδείσων και άλλων ειδών φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ρωτώ γιατί η Ουγγρική κυβέρνηση ανέθεσε σε δύο ε, offshore εταιρείε να ε, πολιτογραφηθούν, τις, ε, τις υιοθέτησε κατά κάποιο τρόπο, τους έδωσε την υπηκότητα. Τι κάνουμε άμα η κυβέρνηση το κάνει αυτό. Και η χαλιβουργία. Η χαλιβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία αλλά αν οι κυβερνήσεις, αν τα κράτη θέλουν να ξεκινήσουν πανεθνικοποίηση αυτών των εταιριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, η Κομισιόν τι θα κάνει. Και έπειτα δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, αλλά και σε άλλους τομείς μπορεί να προκύψει τέτοια κατάσταση, να χρειάζεται να παρέμβει το κράτος. και να λειτουργήσει ως αγοραστής για τις, ε, τους τομείς, για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Κομισιόν τι άποψη έχει. Καταρχάς, για δικαιοδοσίες τρίτων χωρών. Πράγμα το οποίο ήταν προτεραιότητα για πολλά χρόνια. Όταν ήμουν στην ε, ΕΚΟΦΗΝ και προσπαθούσαμε να διαπραγματευτούμε με τρίτες χώρες ώστε να τους, φέρουμε, να τους κάνουμε να κατανοήσουν ε, τι γίνεται για τις κατοικές ενισχύσεις, ε, ε, τις επιδοτήσεις κτλ. Ακόμα και αν δεν ισχύουν τα ίδια πράγματα όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποχρεωνόμαστε από το κοινό νομικό πλαίσιο, έχουμε πολλά κέρδη εάν ε, καταλήξουμε να έχουμε την ίδια ε, αντίληψη. Για παράδειγμα, το Στάν είναι μια χώρα που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για την ε, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, άρα λοιπόν υπόκειται στους κανόνες κρατικών, περικρατικών ενισχύσεων και αυτές ε, τους επιβλέπει η ΕΦΤΑ ως εποπτική αρχή και επιβάλλει ε, ε, τις, τους κανόνες αυτούς. Αυτό είναι ένα είδος επέκτασης των, της, της συνεννόησης και των αντιλήψεων για την Ελβετία. Ε, δεν ισχύουν βέβαια οι, οι δικές μας συνθήκες για τις κατοικές επιδοτήσεις, ωστόσο η συμφωνία που ισχύει είναι παρόμοια με αυτή ε, που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις. Έχουμε δηλαδή κάποιο περιθώριο λιγμό όταν πρόκειται για τρίτες χώρες και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό στο πλαίσιο του ΩΣΑ, ε, του ΠΟΕ και στα διεθνή φόρα, ώστε ε, να υπάρχει όντως πραγματική φορολόγηση ότι τα κέρδη δεν μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη μέσα στην Ευρώπη και μετά εκτός δικαιοδοσίας μας. Τώρα, είμαστε ουδέτεροι όσον αφορά την ιδιοκτησία. Έχουμε τον, τον ίδιους κανόνες, είτε οι επιχειρήσεις είναι ιδιωτικές, είτε είναι κρατικές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε διαφορετικές παραδόσεις στα κρατημέλη. Ορισμένοι έχουν απελευθερώσει πολύ, ενώ άλλα κράτη ε, ακολουθούν την παράδοση των κρατικών εταιριών. Το θέμα είναι να μπορούν να ανταγωνιστούν επίσης όρις στις ίδιες αγορές. Βεβαίως το κράτος μπορεί να ενεργήσει ως επενδυτής. Εξαρτάται μόνο αν ενεργεί ε, με κρατική ενίσχυση, ενώ αν είναι επενδυτής της αγοράς, τότε δεν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι αρκετά ανοιχτή η κατάσταση. Όμως υπάρχει μια ειδική υπόθεση που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί άλλο είναι να έχουμε ισότιμο πεδίο στην Ευρώπη, αλλά το καλό είναι να υπάρχει παγκοσμίω και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε τη διαθεσή μας για να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Για το χάλιβα, η δικιά μου προσωπική αίσθηση είναι ότι πράξαμε το σφάλμα το 2003 να αφήσουμε να πεθάνει η ΕΚΑΧ, που ήταν η πρώτη ιστορικά συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έδινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα να έχει μια πραγματική πολιτική χάλιβα και άνθρακα και βοήθησε κάποιες χώροι μέλη τη δεκαετία του 80 να ε, αλλάξουν. Ήταν βέβαια δύσκολο, τους κόστησε πολύ να κλείσουν κάποια ορυχεία, χαλιβουργία, με βοήθεια όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέποντας να λειτουργήσουν όλα με δικαιοσύνη. 50 χρόνια κράτησε και δεν ανανεώθηκε. Είναι κρίμα. Και είναι ακόμα πιο κρίμα για τη συνθήκη αυτή έδινε στην Ευρώπη φορολογικά έσοδα τα οποία πήγαιναν αμέσω κατευθείαν στον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούσαν τα χρήματα αυτά σε αναδιάρθρωση. Σάτισλαφ Κρασνουντεύσκη τώρα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος ανέφερε τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτρόπου πιο συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει, είναι καλή, γιατί χωρίς τη συνεργασία των χωρών μελών βέβαια δεν μπορείτε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας αποτελεσματικά. Η μία μου ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με τις πληροφορίες που παίρνετε από τις χώρες μέλη όσον αφορά του, τις φορολογικές ρυθμίσεις. Τι πληροφορίες σας σας δίνουν. Γιατί οι χώρες μέλη πράγματι έχουν πολύ διαφορετικές φορολογικές ρυθμίσεις. Υπάρχει το απόρριτο μερικές φορές Και τέτοιες ρυθμίσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται για να κρύβουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε και χωρίς να παραβιάσετε την επικουρικότητα καταφέρνετε να έχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Δεύτερον, η διαδικασία της φοροαποφυγής είναι πολύ προβληματική περίπτωση αυτή. Γιατί υπάρχουν χώρες που από το 89 φτιάχνουν τον καπιταλισμό εκεί. Είναι αλλιώ τα πράγματα στην Ιταλία, στη Γαλλία, που από το 45 οργανώνουν τον καπιταλισμό τους. Για άλλες όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και υπάρχει συμμετοχή πολλών ξένων επιχειρήσεων. Οι ξένες αυτές επιχειρήσεις για χρόνια ήταν προνομιούχες. Και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ο κόσμος το καταλάβαινε, το ήξερε και έλεγε εντάξει είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να έχουμε τη δικιά τους πραγματογνωμοσύνη, για να μας βοηθήσουν τεχνολογικά, ε, στην πληροφορική κτλ. Οι χώρες Ανατολικής ε, λοιπόν ε, Ευρώπης όπως και η δικιά μου η Πολωνία θα θέλαν να βρεθεί και πάλι ισορροπία ανάμεσα στις δικές τους επιχειρήσεις τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και των μεγάλων πολυεθνικών που μας βοήθησαν βέβαια να φτιάξουμε τη δικιά μας οικονομία της αγοράς. Είναι ευρύτερο βέβαια το ζήτημα, είναι κοινωνιολογικό και οικονομικό. Οι χώρες αυτές μπορούν ε, να βασιστούν στη δικιά σας κατανόηση και στήριξη ώστε να καταφέρουν να πετύχουν και πάλι την ισορροπία αυτή στην οποία αναφέρθηκα πριν. Ευχαριστούμε. Η Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση. Η συνεργασία με τις χώρες ε, μέλη. Ναι, υπάρχει συνεργασία. Μερικές φορές βέβαια μας παίρνει λίγο χρόνο να τα καταφέρουμε. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες είναι καλή, αρκετά καλή συνεργασία με τις χώρες μέλη. Φυσικά πρώτα απ' όλα ζητήσαμε κατάλογο με γενικά όλες τις φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν οι χώρες μέλη και μετά ζητήσαμε συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εταιρείε. Και πήραμε τις πληροφορίες αυτές που ζητήσαμε. Βέβαια, όντως υπάρχει το θέμα του απορρίτου μερικές φορές. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες είναι υπό το καθεστώς του απορρίτου και γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγουν από το κτίριο. Γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικά ζητήματα και ρυθμίσεις. Αλλά εμείς βέβαια φροντίζουμε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην χρησιμοποιείται σαν άλλο το απόρριτο. Αλλά η ισορροπία είναι το βασικό. Πώς θα πετύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Για το δεύτερο που είπατε. Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν ίσχυε όμω μόνο για τις νέε χώρες ή μόνο τη Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης που δημιούργησαν τον καπιταλισμό εκεί τι τελευταίες δεκαετίες, ισχύει για όλες τις χώρες, γιατί οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν και αυτές την ίδια ευκαιρία όπως και οι μεγάλες. Οι μεγάλε μπορεί να έχουν περισσότερη δύναμη, να προσφέρουν περισσότερο καπιταλισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι οι μικρές ε, και μεσαίες εθνικές επιχειρήσεις πρέπει να πλήττονται από τις μεγάλες. Ισχύει αυτό λοιπόν σε όλες τις χώρες και κάθε επιχείρηση πρέπει να ξέρει ότι καμία επιχείρηση δεν είναι υπερβολικά μεγάλη για να ξεφεύγει από τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις. Πάντως κάποιες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αλήθεια ότι αποτελούν την ε, σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τις χρειαζόμαστε και εμεί τι χρειαζόμαστε και, αυτέ πρέπει, και αυτές πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε εμά. Ευχαριστώ. Τόρμεντς, εκ μέρου του Άλντε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, που ήρθατε εδώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Μέχρι στιγμή. ξέρουμε λίγα πράγματα για το Panama Leaks, αλλά στην Ζιντο Τσετσάιτουγκ υπάρχει ένα γράφημα Δηλαδή το LuxLeaks ήταν 4 GB ε, και το ParmaLeaks είναι 2,6 TB. Εάν ε, το LuxLeaks σας έδωσε 600 υποθέσεις, τότε εδώ πέρα ε, μετρήστε μόνοι σας ε, πόση δουλειά σας περιμένει. Όπως είπα, λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Διαβάσαμε την Süddeutsche Zeitung και τις δικές μας εφημερίδες, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση περίεργη. Δηλαδή παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι με τις εταιρείε και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα έχουν πει μόνο όσα εξαναγκάστηκαν να πούν. Και μετά την υπόθεση του Παναμά θα πούν «Α, ναι, το είχαμε ξεχάσει και αυτό». αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε δηλαδή. Οπότε οι πληροφορίες ε, τις οποίες λαμβάναμε μέχρι τώρα ίσως να μην ήταν ε, ακριβείς ή ίσως να ήταν πολύ περιορισμένες. Μήπως έπρεπε να ξαναδείτε τις περιπτώσεις που έχετε ήδη κλείσει και να δείτε τι σας είπαν και τι θα έπρεπε να έχουν πει. Μετά, άλλη μία ερώτηση. Είπατε πως αν το παραθυράκι ισχύει για όλους, τότε προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα κάποια από τα παραθυράκια είναι πάρα πολύ ακριβά και εξορισμού, άρα δεν είναι διαθέσιμα για όλους. Και μετά νομίζω πως ο συνάδελφος κ. Κασνοτεύσκη τα είπε σωστά. Στο έργο του Αλεξάνδρ Γκερσέγκο έλεγε ότι οι χώρες οι οποίες ε, ε, ήρθαν πιο μετά στο σύστημα αυτό δεν είχαν ε, χρόνο να οικοδομήσουν τους απαραίτητους οικονομικούς θεσμούς. Έχετε όμως πολλή δουλειά μπροστά σας. Η Επίτροπος. Δεν πρέπει να παραπονιέται κανείς όταν έχει δουλειά. Και βεβαίως, κοιτάξτε, προφανώς τα παραθυράκια, ακόμα και τα παραθυράκια που ισχύουν για όλους είναι πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς και εσείς και το Συμβούλιο περάσατε νομοθεσία για να κλείσουν τα παραθυράκια της ε, νομοθεσίας αποφυγής διπλής ε, φορολογίας που κατέληγε σε διπλή μη φορολογία που ήταν παραθυράκια για όλους αλλά προβληματικά. Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι πως αν ισχύει για όλους δεν είναι κρατικές ενισχύσεις επειδή δεν είναι επιλεκτικά. Και εμείς με τις κρατικές ενισχύσει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλεκτική μεταχείριση. Όταν κάτι ισχύει για όλους είναι μια γενική νομοθεσία. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό ακριβώς εκτιμώ τη δουλειά που έχει γίνει, γιατί πολλά παραθυράκια έχουν κλείσει. Για το θέμα των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Μια που είναι κρατικές ε, ενισχύσεις ε, μιλάμε συχνά με τα κράτη-μέλη. Ε, δεν είμαστε μόνο εμείς οι εθνικές φορολογικές αρχές που ίσως έχουν πρόβλημα εδώ. Ένα από τα ζητήματα που ήταν καλύτερο πριν από χρόνια είναι πως ε, τώρα υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για το προσωπικό εισόδημα και για τα εταιρικά συστήματα. Οπότε δεν μπορεί απλά κανείς να επαναπατρίζει χρήμα σε κάποια ευρωπαϊκή τράπεζα ε, εκτός της χώρας ε, στην οποία είναι φορολογικός κάτοικος χωρίς να είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτό το εισόδημα. Οπότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή η υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχουμε κλείσει και τα έχουμε καταφέρει όλα. Αντιθέτως, αλλά θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερο, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε αποκτήσει την γνώση, ξέρουμε το τι συμβαίνει και βεβαίω παρά το ότι είναι ακόμα νωρί, θεωρώ πως υπάρχει εδώ πέρα ε, ένα κίνητρο για τον νομοθέτη και τις εποπτικές αρχές για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ Φάμπιο Ντεμάζη. Κυρία Βεστάκη, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί, αγόρι, οι γονεί μου μου διάβαζαν ένα παραμύθι που λεγόταν πόσο ωραίος είναι ο Παναμάς. Χτες είδαμε τι ε, άσχημο πρόσωπο του Παναμά, έναν Ρώσο νονό ε, που εμπορεύεται παιδιά, έναν τρομοκράτη, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ε, τον Λιονέλ Μέση, την FIFA και τη σύζυγο του κυρίου Κανιέτη, του συναδέλφου σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, ο Παναμάς δεν είναι πλέον στην ε, γκρίζα λίστα του ΩΣΑ για το ξέπλυμα χρήματος ο λέει ότι ανταλλάζουν καθημερινά δεδομένα, αλλά κοιτάξτε Εγώ πήρε, επικοινώνησα και με την εταιρεία αυτή στον Παναμά και τους ρώτησα αν μπορούν να με βοηθήσουν να βγάλω λεφτά από την Ευρώπη και με διαβέωσαν ότι η κυβέρνηση του Παναμά ποτέ δεν θα ανταλλάξει τέτοιες πληροφορίες. Οπότε, με αυτό το θέμα, όπου βλέπουμε ότι η τωρινή Προεδρία του Συμβουλίου, η Ολλανδία, η οποία έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με τον Παναμά, θεωρώ πως δεν έχει ε, λειτουργήσει αυτό. Με βάση όλα αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα θέλατε να συνεχιστεί αυτή η δουλειά που κάνουμε και αν θα θέλατε να υπάρχει και μια τρίτη θητεία αυτής της Επιτροπής να γίνει μόνιμη. Μετά θα συζητήσετε μετά τον ε, συναδελφό σας, τον κύριο Κανέτε, την περίπτωση αυτή. Τρίτον, έχουμε, θα δείτε την δυνατότητα αφαίρεσης ε, της, ε, λειτουργία, της άδειας λειτουργίας ε, τραπεζών όταν συμπράττουν σε τέτοιες ενέργειες. Και μετά μας είπατε πως οι αναφορές αναχώρα δεν θα αφορούν τους φορολογικούς παραδείσους εκτός Ένωσης. Και η Κομισιόν μας λέει πως αυτό γίνεται για λόγους ανταγωνισμού. η Κομισιόν έκανε ακριβώς το αντίθετο περιέλαβαν ε, και φορολογικούς παραδείσους εκτός Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε την διαφορά μεταξύ Αυστραλίας και Ένωσης. Και τέλος, το τμήμα σας ε, θεωρείτε πως ε, είναι επαρκώς στελεχωμένο για να εφαρμόσει σωστά την νομοθεσία. Η ΕΠΑ παραπονιούνται ότι ασχολείστε επιλεκτικά με εταιρείε και κάποιος από τη δικιά σας την υπηρεσία μας είπε πως δεν έχετε επαρκές προσωπικό για να ασχοληθείτε με όλες τις υποθέσεις. Πολλές ερωτήσεις. Καλές βεβαίως, όλες καλές είναι. Λέει. Κύριος Ντεμάζη. Λοιπόν, ωραία, ε, κοιτάξτε την ερώτηση για το τι θα κάνει η Επιτροπή σας θα την αφήσω στον πρόεδρό σας. Αλλά ελπίζω να συνεχίσετε το έργο σας γιατί θεωρώ πως ε, στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και τις μέρες αυτές Εντάξει, δεν μας προξενεί η έκπληξη ότι ο Πάναμας ε, βρίσκεται στη μαύρη λίστα 8 χωρών, αλλά ε, οπωσδήποτε ο αριθμός των περιπτώσεων προξενεί κάποια έκπληξη. Και άρα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όχι μόνο για τους νομοθέτες, αλλά και για τους ερευνητές στο μέλλον για να δουν ποιο είναι το θέμα. Και οπωσδήποτε και οι επιχειρήσεις να δουν τι είναι το θέμα. Και βεβαίως ε, και οι υπόλοιποι θα το σκεφτούν. Θα λένε θέμε να βρεθούμε στο ίδιο τσουβάλι με αυτούς τους οποίους αναφέρατε εσείς τι θα συμβεί, παραδείγματο χάρη στην εταιρεία μας, στο σήμα μας. Και αυτός είναι ένας καλός λόγος βεβαίως για διαφάνεια. Και δεν είπα τίποτα για το πόσο θα είναι η πρότασή μας όταν θα μπει επιτάπητος ε, στο προσοχές μέλλον. Απλά είπα ότι είναι σημαντικό να σεβόμαστε την δικαιοδοσία και βεβαίως μετά να τα εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο. Και ευχαρίστως να κάνουμε αυτή την συζήτηση όταν θα έχουμε μια πρόταση επιτάπητος. Γιατί νομίζω ότι έχουμε την ίδια οπτική γωνία. Η απάντηση είναι όχι. Λέει ο πρόεδρος. Θα το συζητήσουμε όμως μετά. Για τους πράσινους Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πράγματι, έχουμε χρόνο μπροστά μας να ασχοληθούμε με τον Παναμά. Πάντως, από πλευρά της Ισπανίας σας διαβεβαιώ ότι θα έχουμε πρώτη και παραδείγματα αρκετά για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και στοιχεία που θα συνδέσουν τη χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν, ευχαριστώντας σας για το έργο σας, κυρίως για το LuxLeaks, να σας πω εξής, η ομάδα μας, όπως γνωρίζετε, έχει κάνει τη δικιά της τη μελέτη για το θέμα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις οι φορολογικές αυτές ρυθμίσεις έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις που ελάχιστα δραστηριοποιούνται στην ίδια τη χώρα του Λουξεμβούργου. Προστατεύονται δηλαδή φορολογικά απλώς και μόνο. Ε, πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Αμερική, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Γαλλία και αλλού. Συμφωνείτε με το συμπέρασμα αυτό της δικιάς μας έρευνας και προβληματισμού που συμπληρώνει νομίζω τη δικιά σας. Δεύτερον, αναφερθήκατε στα υπερβολικά κέρδη στο Βέλγιο. Και εμείς είπαμε ότι το βελγικό κράτος πρέπει να πάρετε 700 εκατομμύρια από τις επιχειρήσεις αυτές. Εσείς έχετε νέα από τη βελγική κυβέρνηση από αυτού. Έχετε την επιβεβαίωση ότι το βελγικό κράτος θα πάρει πράγματι τα 707 εκατομμύρια. Θα δημοσιεύσετε το κατάλογο με τις επιχειρήσεις που χρωστούν στη βελγική κυβέρνηση. Γιατί η βελγική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τέτοιο κατάλογο. Και τέλος, ποιο θα είναι το επόμενο δικό σας βήμα αν το Βέλγιο δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του και δεν εισπράξει τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, για να απαντήσει η Επίτροπος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σύμφωνο μαζί σας ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και ότι όντως θα δούμε και την εντολή της Επιτροπής σας για να δούμε πώς μαζί θα, συνεχί... θα συνεργαστούμε στη συνέχεια. Τώρα, για το θέμα αυτό του Βελγίου. Έχει αρχίσει η διαδικασία, αλλά βρίσκεται σε ένα αρχικό στάδιο ακόμα. Υπάρχουν πάνω από 30 περιπτώσεις που πρέπει ακόμα να εξεταστούν για να δούμε ποια είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει να ανακτήσει το Βέλγιο από τις επιχειρήσεις αυτές. Συνεργαζόμαστε με τη βελγική κυβέρνηση για να γίνει αυτό ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πιο περίπλοκο από την Fiat ή την Starbucks και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Τώρα για το ζήτημα της δημοσίευσης των επιχειρήσεων, του ονόματος των επιχειρήσεων, το συζητάμε και αυτό με τη βελική κυβέρνηση. Η δικιά μου η θέση είναι ότι μερικά ονόματα έχουν βγει στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω λοιπόν ότι για κάθε επιχείρηση θα ήταν καλό να ξέρουμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις και ποιες δεν είναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι ύποπτες, ότι μπορεί να βρίσκονται στον κατάλογο. Οπότε είναι κάτι που συζητάμε και εμείς με τις βελικές αρχές. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη δημοψήφιση τέτοιου καταλόγου, αλλά ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε. Όσον αφορά τώρα την ανάκτηση των ποσών, θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Εάν η απόφαση της Επιτροπής δεν τηρηθεί και εφαρμοστεί, τότε θα αρχίσει η διαδικασία επί παραβάση. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του FTD, Μάρκο Τσάνι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για αυτήν ε, την ε, σημερινή συνάντηση. Έχω δύο σειρές από ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τις ε, Ε, το, τις ε, επιχειρήσεις που είναι υπό έρευνα από πλευράς της Κομισιόν. Αναφέρομαι στην ε, Google. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εξετάζει την υπόθεση όσον αφορά τις δραστηριότητες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πιθανή δηλαδή υπόθεση φοροδιαφυγής. Ε, και φόρο αποφυγής. Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι από ότι από το 2014 η Google μετακίνησε τις διεθνείς της ε, δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και από ευρωπαϊκές θηγατρικές 11 δις μέσω μετακίνησης των κερδών στις Βερμούδες, πράγμα που επέτρεψε στην επιχείρηση αυτή να εξοικονομήσει 2 δις σε φόρους. Θέλω να ξέρω αν λαμβάνετε υπόψη αυτού του είδους τους δραστηριότητες και αν κάνετε κάτι για όλα αυτά, αν κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το country by country, την αναχώρα δημόσια έκθεση. Ξέρουμε την εμπειρία των γαλλικών τραπεζών, ορισμένε μάλιστα ήρθαν εδώ σε ακροάσει ενώπιον τη Επιτροπή. μου. Κατά κάποιο τρόπο η αναχώρα έκθεση λειτουργεί. Η Γαλλία, οι Γαλλικέ Τράπεζε ήταν οι πρώτε που δημοσίευσαν αυτού του είδου τα στοιχεία, με ατελή τρόπο βέβαια, αλλά στους ισολογισμούς τους ε, τα παρουσίασαν τα στοιχεία αυτά και κάποιες ε, ε, ενώσεις αποκόμισαν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και θα μπορούσαν αυτές να τις χρησιμοποιήσουν και οι ερευνητικές οι ανακριτικές αρχές για να δούμε τι τρέχει με αυτές τις τράπεζες. Εσείς Ποια γνώμη έχετε σε σχέση με το γεγονός ότι η αναχώρα εκθέσεις για τις τράπεζες θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στο επίπεδο των ομίλων. Πέρα από αυτό που ήταν η πρόταση που είναι επιτάπητος και υποσυζήτηση από πλευρά της Κομισιόν. Και όσον αφορά την υπόθεση του Παναμά, ρόλος των ΙΠΑ. Θυμόμαστε και θυμάστε και την επιστολή που λάβατε για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει υπερβολικό ζήλο ε, στις έρευνες ε, που αναμειγνύονται και οι αμερικανικές εταιρείες. Δεν σας φέρετε λοιπόν παράξενο τα πρώτα νόματα που προέκυψαν από αυτή τη διαρροή δεν υπάρχει ούτε μία αμερικανική εταιρεία, αμερικανός χρηματιστής Ποιο είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι ΙΠΑ δηλαδή μέσα σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής δεδομένης και αυτής της επιστολής κατά τη γνώμη μου ήταν ε, εξαιρετικά ατυχής. Παρακαλώ συνάδελφοι να αποφεύγετε τις πολύ μακρές ερωτήσεις αν θέλετε να λαμβάνετε και ουσιαστικές απαντήσεις γιατί γιατί αν εσείς χρησιμοποιείτε όλο το χρόνο, λέει Επίτροπος, εγώ ξεφεύγω πολύ εύκολα. Τρεις σημαντικές ερωτήσεις θέσατε. Καταρχάς, ήμασταν σε επαφή με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ε, ρύθμιση της υπόθεσης φορολόγησης της Google. Είναι όμως πολύ νωρίς, δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και ε, δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε αυτή την, ε, την έκβαση μάλλον, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Για τι αναχώρα εκθέσει είναι πολύ σημαντικό και είναι η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ε, οι εκθέσει να είναι, οι αναφορέ να είναι τμήμα τη νομοθεσία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση, που όταν αυτή ήταν στο αποκορύφωμά τη και ήταν πάρα πολύ θετική αυτή η προσπάθεια, γιατί αποτέλεσε ένα μοχλό για τη διευκόλυνση ε, μιας πολύ πιο θετικής προσέγγισης από πλευράς των χωρών και για την υπόλοιπη οικονομία και αυτό είναι πολύ θετικό. Νομίζω πως επίσης τα πρώτα χρόνια δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε χώρα να εφαρμόζει ένα ξεκάθαρο σύνολο κανόνων ώστε να μην γίνεται στρεβλωμένη εικόνα της κατάστασης του τομέα. Εδώ ήταν πολύ θετικά τα βήματα πιστεύω και θα βρείτε πως έχοντας το αυτό υπόψη θα περιλαμβάνεται στην πρότασή μας αυτή η δημόσια διαβούλευση των χώρα εκθέσεων. Τώρα, όσον αφορά τη ΣΥΠΑ έχουμε κοινού στόχους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, όσον αφορά τον ΣΑ συμφωνούν μαζί μας, ε, δηλαδή για τη μετακίνηση των κερδών και το βασικό σχέδιο και την έγκριση του G20 και του ΟΣΑ για να προωθηθεί μια συμπεριφορά που θα διευκολύνει την, νομοθ... την φορολόγηση. Εδώ είμαστε μαζί. Προχωράμε παράλληλα. για μια Αμερικανική εταιρεία είναι το ίδιο σημαντικό οι ανταγωνιστές τους στην Ευρώπη να μην έχουν ε, πλεονεκτήματα. Δεν είναι θέμα προκατάληψης. Ε, ε, γιατί αν υπάρχει ειδικά πλεονεκτήματα για οποιαδήποτε εταιρεία, την αμερικανική ή την ευρωπαϊκή, αυτό είναι πρόβλημα. Ε, πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Έχουμε λάβει ένα σωρό αποφάσει τα τελευταία χρόνια για ανάκτηση και μόνο μια χούφτα ήταν αμερικανικές εταιρείες. Κατά τα λοιπά, ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κρατούν ε, τη suspense ε, για... θα ήταν εντυπωσιακό να μην υπάρχουν Αμερικανοί αμερικανικά συμφέροντα μέσα, στο, με, μέσα στο χαρτιό του Παναμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα του Ισπανού συναδέλφου για το Βέλγιο. Μας είπατε πως θα έχετε μια καλή συνεργασία, όμως τα πράγματα στο Βέλγιο ακούγονται κάπως διαφορετικά. Ο Υπουργό Οικονομικών λέει πω θα ασκήσει έφεση στην απόφασή σα ο κύριος Φανόβερφελντ, ο οποίος παρετήθηκε από συναδελφό σα για να αναλάβει το Υπουργείο. Και το ΕΝΒΑ, το μεγαλύτερο κόμμα της κυβέρνησης, είπε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο του Βελγίου πως πρόκειται για τρέλα όταν μιλάμε για μέτρα κατά του Βελγίου και πως πρόκειται για μια παράνομη επίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο βελγικό φορολογικό σύστημα. Ο κύριος Φαν Όβερφελτ, ο υπουργό Οικονομικών, αυτά. Και λέει πως... Ε, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επανέλθουν σε μια μαλλότητα. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, ό,τι είναι αναγκαίο για να λάβουν χώρα οι πληρωμές. Και ο εκπρόσωπο του προσέθεσε πως οι αποφάσεις αυτές ε, δεν ήταν σωστές και αναρωτιέται ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά την ε, έφεση αυτή. Και αναρωτιέται λοιπόν κανείς ε, ποιο είναι το σχέδιό σας σε σχέση με το Βέλγιο. Γιατί αυτό το οποίο λέτε Ακούγεται θετικό, αλλά η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική και η πολιτική επικοινωνία στο Βέλγιο, στο κοινοβούλιο είναι ε, κάπως διαφορετική με... Ε, από αυτό το οποίο μας λέτε εσείς. Δεν είναι αυτό το οποίο μας είπατε εσείς ε, καθόλου. Και η δεύτερη ερώτηση θα γίνει, θα ασχολείστε μόνο με μικρά κράτη-μέλη ή θα δείτε με το τι κάνουν και χώρες μεγαλύτερες από το Βέλγιο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σύμφωνα με την ε, εμπειρία μου, μπορεί κανείς να συνεργάζεται χωρίς να συμφωνεί. Γίνονται νομίζω αυτά. Και βεβαίω μπορεί να διαφωνούμε και να ζητήσουμε από τα δικαστήρια να κρίνουν τούτων λεχθέντων. Η έφεση στις αποφάσεις της ε, Κομισιόν δεν θα σταματήσει τη διαδικασία ανάκτησης ε, των χρημάτων. Αυτή θα συνεχιστεί κανονικά, γι' αυτό ακριβώς συνεργαζόμαστε με τις βελγικές αρχές, όπως ε, για να γίνει ανάκτηση, όπως έγινε και στο Λουξεμβούργο, όπου η φορολογία της Fiat βρίσκεται σε ένα λογαριασμό με τρίτη εγγυητή. Η διαδικασία συνεχίζεται, αλλά ε, δεν υπάρχει πλέον αναταραχή στις αγορές. Και νομίζω πως είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος αυτός. Δηλαδή να μην υπάρχει αναταραχή στις αγορές, να πηγαίνουμε μετά στα δικαστήρια και να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις ε, συνεργασίας. Θα, για το χρόνο δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα δικαστήρια το πόσο γρήγορα θα κινηθούν. Προφανώς ελπίζω να κινηθούν γρήγορα γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα γιατί υπάρχουν σημαντικά διδάγματα μετά για τα κράτη-μέλη για το θέμα μεγάλων και μικρών κρατών μελών. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, ε, κοιτάμε όλα τα κράτη-μέλη και είδαμε ότι κάποια δεν κάνουν καθόλου τέτοιες ε, αποφάσεις. κρατημέλη ακολουθούν τους κανόνες και σε καποια κρατημέλη βρήκαμε φορολογικές αποφάσεις που γύρουν ανησυχίες. Και η ανησυχία μας δεν πηγαίνει με το μέγεθος της χώρας, εξαρτάται από την φορολογική απόφαση. Και νομίζω αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστώ. Αυτό. Κοιτάξτε, εν γέννη πρόκειται για μεγάλες εταιρείες μεγάλων κρατών μελών. που είναι σε στενή επαφή με τα πιο μικρά κράτη-μέλη για να αποκομίσουν συμφέρουσες συμφωνίες. Ανδρέας Βάμπα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε, Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχουν ακουστεί ήδη τα πράγματα, από θα ήθελα εγώ να θέσω ένα διαφορετικό ερώτημα. Είπατε στην εισαγωγή σας πως πρόκειται για νομολογία η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πως υπάρχει νομολογία η οποία λέει πως τα ζητήματα τα φορολογικά πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως και οι κρατικές ενισχύσεις και άρα είστε πολύ αισιόδοξη πως θα προκύψει κάτι από την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου. Εμείς βεβαίω μπορούμε να σας ρωτήσουμε πολύ πιο άμεσα στην Επιτροπή μας γιατί οι διαδικασίες είναι παρόμοιες ε, με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Τι σας κάνει τόσο αισιόδοξη όταν τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται για το ότι θα έχουμε καλύτερη φορολογική συνεργασία τα επόμενα έτη, γιατί τα πράγματα νομικά είναι όπως είναι. Και δεν ε, είναι καλό να κάνουμε εικασίες. Αν, υπάρχουν, αν υπάρχει λόγος αισιοδοξία πρέπει να τεκμηριώνεται το δεύτερο ερώτημα. Ε, χρησιμοποιείται πάντα διεθνείς αρχές, ε, όπως αυτό το Arm's Length Principle και τώρα και η Κομισιόν έχει κάποιες επιφυλάξεις για το εάν αυτές οι πολύ γενικές ε, αρχές ε, μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται γιατί αφήνουν πάρα πολλά περιθώρια ερμηνείας ε, και διακριτικής ευχέρειας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτό. Σας ευχαριστώ, η κυρία Επίτροπος. Οι αρχές του ΩΣΑ και είναι πολλές οι αρχές, δεν είναι μία. Λένε πως υπάρχει ε, υποχρέωση βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε την αρχή που ισχύει στην περίπτωσή μας, όχι αυτή που μας βολεύει. Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει περιθώριο για έλεγχο ε, των ε, κρατικών ενισχύσεων μετά, εφόσον ισχύουν οι αρχές του ΩΣΑ σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε την μέθοδο που αντικατοπτρίζει την ε, πραγματικότητα των αγορών και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για το θέμα της αισιοδοξία τώρα. Πάντα προσπαθώ να το αντισταθμίσω αυτό αλλά κάποια πράγματα νομίζω μας πηγαίνουν προς, δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η δημόσια συζήτηση περί που είναι νομίζω πολύ σημαντική γιατί τίποτα δεν κινητοποιεί τις ε, κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις όσο το να κάνουν ερωτήσεις οι ψηφοφόροι και οι πελάτες τους. Γι' αυτό είναι νομίζω σημαντικό. Και έχει θετική και αυτή είναι και η θετική πτυχή των Panama Papers, ότι επανήλθε το ζήτημα. Δεύτερον, νομίζω πως έχουμε δει αλλαγή, πραγματική αλλαγή. Έχουμε δει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που πέρασαν ε, νομοθεσία πάρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Όταν η Δανία είχε την ε, Προεδρία προσπαθήσαμε να περάσουμε πάλι κάποιες από αυτές τις προτάσεις και κάποιος μου είχε πει ότι ξέχασέ το. Γιατί η δικιά τους η λογική ήταν τώρα η μόδα και δεν επρόκειτο να αλλάξει. Και όμως άλλαξε. Και την υπερψήφισαν κιόλα οι ίδιοι. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν. Ένα από τα πράγματα που διάβασα για το Panama Papers είναι πρακτικά από συνεδριάσεις σε τράπεζες που λένε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η offshore είναι πλέον αδιέξοδο και πρέπει και πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε και οι κοινικοί πλέον πρέπει να ζυγίσουν το ρίσκο του να βλαφτεί η εικόνα, της εταιρείας, η εικόνα της εταιρείας. Ε, ως αντιστάθμισμα της μείωσης της φορολογίας. Έχουμε λοιπόν κάποια πράγματα, κάποιες προϋποθέσεις πραγματικής αλλαγής και ειδικά αν συνεχιστεί η δουλειά του Κοινοβουλίου, νομίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι. Ίσως όχι αύριο ή του χρόνου, αλλά θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Γκόμες, τώρα από τους σοσιαλιστές. Όντως, τα έγγραφα αυτά του Παναμά δεν θα φέρουν τίποτα καινούριο πέρα από τα ονόματα των επιχειρήσεων ή των ατόμων. Υπήρχε το LuxLeaks, η λίστα Λαγκάρντα και άλλα. Οπότε η ερώτηση μου είναι, μπορείτε να βρείτε τι έχει κάνει η Επιτροπή. Γιατί εδώ και καιρό ζητά από τις δικές μου τις αρχές να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία από το Λίχνεστάν και την λίστα Λαγκάρ, αλλά οι αρχές δεν κάνουν τίποτα. Δεν έχουν δημοσιευτεί καν οι κατάλογοι αυτοί. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν μέρος της Τρόικα, που πήρε τόσα εκατομμύρια ευρώ από τις μοσίους υπαλλήλου, από τους συνταξιούχους με το μνημόνιο. Και η κυβέρνησή μας τι έκανε, έδινε φορολογικές απαλλαγές και δεν ενδιαφέρθηκε με όσους συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο Λαγκάρτ. Το έχω ρωτήσει ξανά και ξανά την Επιτροπή και σας έχω ρωτήσει να μου πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει ότι οι χώρες μέλη θα αναλάβουν δράση για τέτοιου είδους ε, σκάνδαλα που αποκαλύπτονται όπως τώρα με τα έγγραφα Παναμά. Η χώρα μου, η Πορτογαλία, είναι μεταξύ των 23 χωρών που έχουν τέτοιες πρακτικές φορολογικών ρυθμίσεων, εντελώς μυστικά βέβαια. Και υπάρχουν και offshore. Το αναγνωρίζω δηλαδή και σας ευχαριστώ που αντιδράσατε στα αυτά που σας έχω γράψει εγώ, αλλά απάντηση πήρατε από τις πορτογαλικές αρχές και για τις κρατικές επιδοτήσεις. Υπάρχει κάποια διαφορά με τη σημερινή κυβέρνηση. Η προηγούμενη δεν είχε απαντήσει σε τίποτα. Η καινούρια αντέδρασε καθόλου. Τέλος για την Apple. Υπάρχουν πληροφορίε ότι συναντηθήκατε με τον κύριο Τιμ Κόξ στις 21 Ιανουαρίου. Το επιβεβαιώσατε κι εσείς. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Apple. γιατί ο Τιμ Κόξ ήθελε να μιλήσει μαζί σας. απάριτο; Εμπίπτει στο απόρριτο. Λοιπόν, παρακαλώ, απάντηση. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση είναι δύσκολη για μένα. Δύσκολο να απαντήσω, γιατί είναι δύσκολο να συγκρίνω ποια ήταν η κατάσταση πριν και ποια είναι η σημερινή προσέγγιση. Είναι δύσκολο να κάνω αυτή τη σύγκριση. Μέχρι τώρα Έχουμε λάβει υπόψη μας από διαρροές, από πληροφορίες, έχουμε συσσωρεύσει ό,τι πληροφορίες μπορέσαμε να έχουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε για την έρευνά μας. Γνωρίζοντας βέβαια που αρχίζει η δικιά μας η αρμοδιότητα, αλλά και που σταματάει αυτή για θέματα που είναι παράνομα βάσει του εθνικού ποινικού δικαίου, πρέπει να ερευνώνται από τις εθνικές αρχές ή από την αστυνομία σε συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχω πληροφορίες για την Πορτογαλία όσον αφορά το ερωτηματολόγιο μας προς όλες τις χώρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ξέρω να μην μας ενημέρωσαν για αυτά που τους ζητήσαμε να μας ενημερώσουν και για τον κατάλογο δηλαδή των ε, γενικών φορολογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Πορτογαλία, είτε ειδικότερα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Όπως είπε και ο πρόεδρος, οι συναντήσεις είναι ιδιωτικού επίπεδου. Γενικά πάντως, όταν πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις, αυτό είναι ένα θέμα απόλυτα ξεκάθαρο. Έχουμε να κάνουμε με τη χώρα μέλος και αξιολογούμε κατά πόσο η χώρα μέλος αυτή δίνει επιλεκτικά πλεονεκτήματα. Μερικές φορές μιλάμε με τις επιχειρήσεις για να έχουμε πληροφορίες προκειμένου να τους δοθεί ευκαιρία να απαντήσουν, να πούνε κατά πόσο οι πληροφορίες που έχουμε εμεί στη διάθεσή μας είναι σωστές ή δεν είναι. Αν όμως διαπιστώσουμε ότι μια χώρα παράνομα έχει προσφέρει επιλεκτικά τέτοια πλεονεκτήματα, τότε ζητούμε να ανακταθούν τα ποσά από τα πλεονεκτήματα αυτά. Είναι μαθηματικά. Ε, φυσικά μπορεί να παίξει λίγο το ποια χρονιά ξεκίνησε αυτή η ρύθμιση, αλλά γενικά είναι θέμα του κράτους μέλους να υπολογίσει ποιο ήταν αυτό το επιλεκτικό πλεονέκτημα, πόσο κόστιστε και να ανακτήσουν τα ποσά. Κούνα Χούκμαρ. Χόκμαρ, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που έχουμε εδώ σήμερα. Τα σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 2,3 τεραμπάιτ και 11 εκατομμύρια gigabyte. Ε, Η διαφορά είναι μεγάλη. Όταν συζητάμε για την περίπτωση του Παναμά, βλέπουμε ότι είναι ένα πιο ευρύ φάσμα αυτό για το οποίο μιλάμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα για εσωτερική τιμολόγηση των ε, ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων που μπορεί να είναι κάτι νόμιμο, αποδεκτό, τέλος πάντων, και είναι κάτι εντελώ διαφορετικό η νομοποίηση παράνομου χρήματος. Μακριά, κάπου που μπορεί να οδηγεί και σε εξοπλισμού στη Συρία. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Κάποια από αυτά τα ζητήματα είναι παράνομα ως έχουν και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από θεσμούς, νόμιμους θεσμούς που υπάρχουν. Και κάποια είναι εθνικά ζητήματα. Κάποια άλλα απαιτούν μια πιο συλλογική παγκόσμια αντιμετώπιση. Γιατί αν στην Ευρώπη τα χειριζόμαστε με έναν τρόπο στην Αμερική, την Κίνα ή τη Ρωσία με διαφορετικό τρόπο, καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχουν τέτοια κενά που θα μπορούν οι εγκληματίες να χρησιμοποιούν και οι κακοί πάντα θα κάνουν τη δουλειά τους. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους εγκληματίες, δεν βοηθάει πάντα να έχουμε καινούριου νόμους, εκείνοι έτσι κι δεν θα του τηρούν τους νόμους. Φτιάχνουμε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι τελικά πολύ βαρύ για τις επιχειρήσεις οι οποίες δρούν νόμιμα. Γι' αυτό θα ήθελα να το σκεφτείτε λιγάκι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι όλοι μπερδεμένοι σε όλα και το κάθε φαινόμενο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εκεί που ανήκει. Να υπάρξει μια καλή διάρθρωση σε όλα αυτά και πώς θα φροντίσουμε ο σωστό θεσμό να ασχολείται με αυτό που τον αφορά. Και έπειτα, για τι ε, έρευνε και όσον αφορά την Gazprom, με τα στοιχεία που βγαίνουν σιγά σιγά από το Panama Papers, πώς βλέπετε την νομιμότητα της Gazprom. Η Επίτροπος. Το τελευταίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν το ξέρω. Δεν ξέρω την απάντηση. Δεν γνωρίζω ποια είναι η απάντηση στην ερώτησή σας αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια αυτό που λέτε και γιατί και εμείς περιμένουμε πολλά από το έργο της δικιάς σας αυτής της Επιτροπής. Ακριβώς αυτό θέλουμε, να ξεκαθαριστούν τα πράγματα και να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Συστήματος και τι μπορούμε να κάνουμε συνεργαζόμενοι με άλλες δικαιοδοσίες, με διεθνή φόρα. Αυτό είναι το κλειδί για να πετύχουμε αλλαγές. Και προκειμένου επίσης να ξέρουμε ότι είναι παράνομο, προφανές, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, να γίνεται δουλειά από πλευρά τη αστυνομία και συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών για να έχουμε εκεί αποτελέσματα. Αν κάποιος θέλει να κάνει παράνομα δουλειά, ε, εντάξει, θα περάσει στην επόμενη ώρα για να κάνει την παράνομη δουλειά του. Το θέμα είναι όμως να τους δυσκολέψουμε. Η νομοθεσία που πέρασε πριν από λίγα χρόνια πέρασε επειδή δεν υπήρχε αυτόματη ενημέρωση των χωρών μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε. Διότι αναγκαστικά θα ενημερώνουν και οι επιχειρήσεις στις χώρες τους και θα αναγκαστούν να κάνουν και ακόμα περισσότερα. Αυτό λοιπόν που βοηθάει είναι ότι και ο κόσμος σκέφτεται «Μα έτσι θέλω να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, έτσι στα κρυφά και παράνομα» και σιγά σιγά αλλάζει η νοοτροπία. Θα πάρει χρόνο. Όπως είπατε, όντως πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι, να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εξετάζουμε και τι είναι αυτό που πολεμάμε και τότε θα υπάρξει αλλαγή και πρόοδος. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ζητήσω από τους εισηγητές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους μετά από αυτή τη συζήτηση. Τώρα, θέλω να σας πω το εξή, κυρία μου, από τις διάφορες πληροφορίες που μας δώσατε, εγώ κρατάω ότι σκοπεύετε να οργανώσετε συνάντηση εργασίας με τους υψηλά εστάμενους αξιωματούχους στα φορολογικά ζητήματα τον Ιούνιο για να κάνετε έναν απολογισμό από τα συμπεράσματά σας δηλαδή, στο οποίο καταλήξατε μετά από τις έρευνές σας εκατοντάδες τέτοιες φορολογικές ρυθμίσεις. Αν είχαμε το πρώτο σχέδιο συμπερασμάτων νωρίτερα, θα ήταν πολύ καλό να το είχαν οι εισηγητές. Λοιπόν, ο Γέπε. Ναι. Και Εξ ονόματος ε, των ε, δύο εισηγητών σας ευχαριστώ κυρία Βεστάγκερ για αυτή την συζήτηση και για την χρήσιμη νομίζω ανταλλαγή απόψεων και όπως είπε και ο πρόεδρος θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχετε κάνει για το transfer pricing και τις συμφωνίες ε, τιμολόγησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει το αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των εταιριών τα οποία κοιτάτε, κάποια κοινά χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει. Κάποια δομή, κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί. Και επίσης ε, ε, οι χώρες αν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτά αναζητούμε και σε εταιρείε και σε χώρες που έχουν μεγάλη ευθύνη θέλω να πω ότι πριν από 15 μέρες κάποιες από τις μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης ήρθαν εδώ σε μια κρόαση και τώρα ξέρετε πως πρέπει να υποβάλουν δημόσιες αναφορές αναχώρα και ήταν υπέρ για την ε, δικιά τους την ε, καλύτερη λειτουργία και νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο αυτό και εντός και εκτός Ευρώπης και τρίτον όπως ανέφεραν κάποιοι, η συζήτηση για την ανάκτηση. Όταν ε, λαμβάνεται μία απόφαση για ανάκτηση, όπως π.χ. στο Βέλγιο, ξέρετε πως στην έκθεση τάξε, της τάξε 1 υπάρχει μία σύσταση ότι δεν πρέπει να ανταμείβουμε τις χώρες που έκαναν μία παράνομη φορολογική συμφωνία με το να λαμβάνουν και όλα στα λεφτά του φόρου εκ των υστέρων. Δεν είναι και πολύ δίκαιο. Δεν ξέρω λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε για να υπάρχει μια συνέπεια και για τις εταιρείες αλλά και για τις χώρες που ε, συνάπτουν τέτοιες παράνομες ε, φορολογικές ε, συμφωνίες. Δεν μπορεί η τιμωρία του να είναι ότι θα λάβουν και όλα τα χρήματα. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Επιτροπέ. Μια σκέψη για την ανάκτηση. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός να υπάρχει δηλαδή αυτή η ανάκτηση για να έχουν οι επιχειρήσεις ίσως όρους ανταγωνισμού. Και το είπε ο κύριος Άνεμαν ότι ο Βέλγος ε, Υπουργό Οικονομικών δεν θέλει τόσο πολύ να λάβει το δώρο αυτό που θέλετε. Πάει στα δικαστήρια για να μην πάρει τα λεφτά πίσω. Νομίζω λοιπόν πως ε, ένα κράτος μέλος το οποίο έχει μια τέτοια σχέση με μια εταιρεία θα πρέπει να δούμε το τι είναι διατεθειμένο να κάνει. Όσον αφορά την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων. Και βεβαίω το θέμα είναι μετά ε, σοβαρότερο από ένα θέμα ανταγωνισμού γιατί γίνεται θέμα της συνθήκης. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε ακριβώς το να ανακύψουν τέτοιες υποθέσεις. Αυτό είναι ακριβώς ένα ζήτημα κατευθυντηρίων γραμμών και καθοδήγησης. Τι νομίζω πως συμφωνούμε σε πολλά πράγματα και με τον πρόεδρο και τους συζητητές. Ένα πράγμα το οποίο έχω δει είναι πως ε, αν υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ των εταιριών και χωρών που, για τις οποίες ανησυχούμε ότι έχουν κάποια αθέμητα πλέον εκτήματα είναι ότι απλά θέλουν να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Αλλιώς είναι από όλους τους κλάδους, είναι μεγάλες εταιρείες, κάποιες είναι πολύ πιο μεγάλες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι ζήτημα κλαδικό που περιορίζεται σε έναν κλάδο, απλά θέλουν να πληρώσουν λιγότερους φόρους. αλλά θα επανέλθουμε και θα αναζητήσουμε αυτά τα οποία λέτε. Ε, λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε εμείς κοινό στοιχείο λοιπόν είναι ότι έχουμε τον ίδιο στόχο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ένας λόγος αισιοδοξία, που, το ερώτημα που έθεσε ο Ανδρέας Φαμ που έφυγε μεταξύ, είναι ότι εάν σήμερα μετά το LuxLeaks και τα Panama Papers Καμία παγκόσμια εταιρεία πλέον δεν έχει την πολυτέλεια να της βγει το όνομα όσον αφορά τους φόρους. Π.χ. για τα smartphone. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες, Όλοι τις ξέρετε, δεν θα τις πω. Εάν μία από τις δύο βγάλει κακό όνομα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και η άλλη καλό, φαντάζεστε. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι ένας λόγος αισιοδοξίας, αλλά βεβαίως έχουμε και άλλους λόγους. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Επίτροπε. Ας μείνουμε λοιπόν σε στενή επαφή για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και κρίσεις για τα διδάγματα που θα πρέπει να αποκομίσουμε από τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει, τις έρευνες που έχετε ξεκινήσει και φυσικά σε σχέση με τα έρφα του Παναμά και τις άλλες αποκαλύψεις του τύπου. Διακόπτουμε για δύο λεπτά τη συνεδρίαση για να συνοδεύσω την κυρία Επίτροπο και να ζητήσω τους εκπροσώπους των τραπεζών να ε, πάρουν θέσεις στην πρώτη σειρά εδράνων.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 Ευχαριστώ που ησυχάσατε. Να δώσουμε πρώτο το λόγο στην κυρία Μπριζίτη Μπόμο, που είναι διευθύντρια του στο τμήμα φορολογία τη Deutsche Bank. Σα ευχαριστώ. Και μετά έχουμε τον κύριο Γκράντα Τζέμισον, που είναι διευθυντή ε, διεθνούς... στο τμήμα διεθνού φορολογία τη Bank of Scotland, τη Τράπεζα Σκοτία. Σα ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Θα ήθελα να πω στου δύο προσκεκλημένους μας ότι η επιλογή των τραπεζών που αποφασίσαμε να καλέσουμε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων γίνεται, έγινε μάλλον σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται με το μέγεθος των τραπεζών ώστε ε, και φροντίσαμε ώστε το πάνελ που καλούμε να αντιπροσωπεύει τις περισσότερες μεγάλες χώρες της Ένωσης. Χάρη στο μέγεθος της τράπεζας λοιπόν που αντιπροσωπεύουν, ε, έχουν ε, σήμερα προσκληθεί εδώ, αν και μάθαμε από τους Financial Times σήμερα το πρωί ότι η Deutsche Bank δεν ήταν πια πρώτη στον κόσμο, αλλά πέμπτη. Πριν από εσά Είχαμε ακροάσει με την HSBC, την BNP Paribas, την Credit Agricole, ING, Unicredit, Santander, Nordea και UBS. Και σήμερα θέλουμε να ακούσουμε και εσάς, γιατί από ό,τι είχαμε καταλάβει, οι προηγούμενες ημερομηνίες δεν σας τέριαζαν. Ε, θα κάνουμε λοιπόν μαζί σας ό,τι κάνουμε και με τις άλλες τράπεζες. Δηλαδή, μετά από μια εισήγηση πεντά λεπτή, από καθένα σας. Θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των ομάδων, δηλαδή σε 12 από τα μέλη μας και, ανάλογα, και σύμφωνα μάλλον με την παράδοσή μας, αν η παρέμβαση των μελών αφορά μόνο μία τράπεζα, θα εφαρμόσουμε το μέθοδο όπως χρησιμοποιήσαμε και με την κυρία Φεστάγια, δηλαδή μία πεντάλεπτη χρονοθυρίδα για την ερώτηση και για την απάντηση, ενώ εάν ο, ο ερωτών θέλει να ρωτήσει και τις δύο τράπεζες θέτοντας διαφορετικές ερωτήσεις στην καθεμιά ή την ίδια και προς τις δύο αλλά επιθυμεί απάντηση και από τις δύο για την ίδια ερώτηση, τότε θα έχουμε χρονοθυρίδες τρίλεπτες. Και σα ζητώ λοιπόν ένα από του ερωτώντε να περιορίσετε τι ερωτήσεις στο ένα λεπτό, ώστε οι προσκεκλημένοι μα να έχουν ένα δίλεπτο για να απαντήσουν. Και ξεκινούμε λοιπόν αυτή την ε, υπόθεση με εσά, κυρία Μπόμα. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι για την συζήτηση για τα επίκαιρα θέματα, όπως φορολογική η και η Μπεύση. Μπριγκίτε Μπον λέγομαι. Εδώ και τέσσερα χρόνια είμαι υπεύθυνη για την παγκόσμια φορολογική λειτουργία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη. Τώρα θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα αγγλικά. Ελπίζω να μην έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την Deutsche Bank πριν αναφερθώ στο ρόλο μου. Ως μια ευρωπαϊκή καθολική τράπεζα, όχι πλέον η νούμερο ένα, Είμαστε μια τράπεζα μέτρα στην Φραγκφούρτη, λειτουργούμε σε 70 χώρες και έχουμε έναν άλλο αριθμό θυγατρικών. Παρέχουμε υπηρεσίες λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής διαχείρισης πλούτου, private banking και βεβαίως trading. Περνάμε αυτή τη στιγμή μια περίοδο αλλαγής και βρισκόμαστε στην φάση εκτέλεση στρατηγικής μας για το 2020. Σκοπεύουμε η τράπεζα να γίνει απλούστερη, πιο αποτελεσματική, εστιάζοντα σε τράπεζες, προϊόντα και πελάτες όπου είμαστε πιο ισχυροί. Σκοπεύουμε να γίνουμε λιγότερο επιρρεπεί στον ε, κίνδυνο, αποσυρώμενοι από κάποιες ε, σχέσεις ε, εταιρικές και να είμαστε πιο πειθαρχημένοι. Οι διαδικασίες για να γνωρίζουμε τους πελάτες μας έχουν ενισχυθεί και λαμβάνουν υπόψη και τις φορολογικές διαδικασίες. Έχουμε ένα εύρωστο σύστημα καταπολέμησης του ξεπλήματο χρήματο σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και το δίκαιο των άλλων χωρών όπου λειτουργούμε. Λαμβάνουμε πολλέ δραστηριότητε για να ενισχύσουμε του ελέγχου αυτού. Οι υπάλληλοι τη τράπεζα έχουν ξεκάθαρε οδηγίε μέσω ενό κώδικα συμπεριφορά για το πώ θα πρέπει να λειτουργούν ε, για λογαριασμό τη τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένε αξίε και πιστεύω, οι οποίε περιλαμβάνουν την ακαιρεότητα, την βιώσιμη απόδοση, την καινοτομία, την πειθαρχία και την συνεργασία. Ο κώδικας τονίζει τον ρόλο της ε, τράπεζας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και στην ανείχνευση και καταπολέμηση ανήθικων εταιρικών πρακτικών. Επίσης, ε, λαμβάνουμε υπόψη τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών μας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στον ρόλο που παίζει το τμήμα το φορολογικό της τράπεζας. Πρώτα απ' όλα, στόχο έχουμε την συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και τις υποχρέωσεις μας. Φροντίζουμε η τράπεζα να πληρώνει τους φόρους που της αναλογούν. Δεύτερον, εγκρίνουμε προϊόντα και συναλλαγές που κάνει η τράπεζα ε, για να δούμε εάν συμμορφώνονται με την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Δεν δίνουμε φορολογικές συμβουλές σε πελάτες, όμως ε, φροντίζουμε όταν υπάρχουν κάποιες πρακτικές αυτές να γίνονται για επιχειρηματικούς λόγους. Έχουμε λοιπόν κάποιες αρχές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας πέραν από το ότι τονίζουμε την αναγκητή συμμόρφωση ε, με την φορολογική νομοθεσία, τονίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το πνεύμα και η πρόθεση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς ε, διακυβεύεται το κύρος ε, της τράπεζας και η σχέση της με τους πελάτες, της, τους πολιτικούς και τις ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τα κράτη και τις φορολογικές αρχές με έναν τρόπο ο οποίος εστιάζει κυρίως στην πρόληψη και την συνεργασία. Εδώ πέρα τελειώνει αυτή και είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ντάνκισον, κυρία μου. Δίνω τώρα τον λόγο στον κύριο Τζέιμσον. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Γκρόντο Τζέιμσον και είμαι επικεφαλής στο τμήμα της φορολογίας της ε, Τράπεζας της και είμαι σήμερα εδώ μαζί με τον κύριο Τόρσμα που είναι επικεφαλή του Τμήματο Διεθνού φορολογία. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο και εκτιμούμε την πρόσκληση εδώ, καθώς και τη σημασία των ζητημάτων στα οποία εστιάζεται η Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας, κάνω μια σύντομη, να σας δώσω μια σύντομη εικόνα και τέλος να κάνω κάποια σχόλια για τα ειδικά θέματα φορολογίας που εξετάζει η Επιτροπή σας. Καταρχά, η γενική εικόνα. Η Τράπεζα τη Σκοτία ε, έχει υποστεί τεράστιε αλλαγέ την τελευταία δεκαετία μετά από μια περίοδο μεγάλη ανάπτυξη ε, συμπεριλαμβανομένη ε, τη αγορά ενό μεγάλου τμήματο τη IBM AMRO, τη χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων τη Βρετανία. Υπήρξε μια θεμελιώδη αλλαγή στην οτροπία και στον εστιασμό. Έχουμε διάφορα franchises και ο πυρήνα των εργασιών μα εστιάζεται στον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η στρατηγική είναι να είμαστε ισχυρότεροι, πιο απλοί και δικαιότεροι. τράπεζα, για, δηλαδή να κάνουμε λιγότερα πράγματα, αλλά να τα κάνουμε καλά όσον αφορά το, και το, τους νόμους, την, το κίνδυνο, και ο πελάτη είναι στο επίκεντρο των όσων κάνουμε. Το 2015 πάνω από το 85% των κερδών ε, γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 70 εκατομμύρια ε, ιδιώτε, αλλά και επιχειρήσεις ε, εξυπηρετήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά την πορεία μα από μια παγκόσμια τράπεζα σε μια απλούστερη, μάλλον οργανισμό που βασίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε αναδιαρθρωθεί τα τελευταία χρόνια Έχουμε περιορίσει το, διεθνή μας, το διεθνές, μα, διεθνές μας αποτύπωμα και έχουμε ενισχύσει την ε, κεφαλακή μας θέση. Ως με της μεταρρύθμισης μια, υπάρχει ένα μεγάλο project για ορθολογισμό. Το 2008 μετά από την αγορά ενός τμήματος της IBM AMRO έχουμε αποκτήσει έτσι πάνω από 2.000 θηγατρικές εταιρείε και το 2015 είχαμε περιορίσει αυτόν τον αριθμό στις 800 και εργαζόμαστε για να τι περιορίσουμε ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά την φορολογική στρατηγική μα, εμεί διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τι φορολογικέ ρυθμίσει κάθε χώρα με τι οποίε συνεργαζόμαστε ε, και ακολουθούμε τον κώδικα πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2009, πράγμα το οποίο μα οδηγεί όχι μόνο στο πνεύμα αλλά και στην πράξη σε ανοιχτή και επικοδομητική σχέση με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, εμείς ε, διεπόμεθε από τους γενικούς κανόνες της Βρετανίας. Δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία ε, συμφωνία που προσπαθεί να με στόχο την αποφυγή φορολόγησης είτε για μας είτε για κάποιον πελάτη μας. Ε, και μάλιστα αντιθέτως έχουμε θεσπίσει πολύ ισχυρούς κανόνες και ελέγχους ώστε να το αποφεύγουμε αυτό. Επίσης δεν πρόκειται να προβούμε σε τεχνητές ε, ε, ε, συναλλαγές πάλι με στόχο την φοροδιαφυγή ή την φοροαποφυγή. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στις ευθύνε μας υπό την ΦΑΤΚΑ και υπό το, τα, τις προδιαγραφές του ΩΣΑ για κοινέ ε, τις κοινές προδιαγραφές μάλλον για τις εκθέσεις υπό τον ΩΣΑ. Αν και όπως είπα περιοριζόμαστε περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξεκολουθούμε να έχουμε δραστηριότητες ε, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου με, διάφορα, με χώρες με διάφορα επίπεδα φορολόγησης. Δεν χρησιμοποιούμε όμως αυτές τις ε, ε, δικαιοδοσίε Χαμηλή φορολογίας για να αποφύγουμε τη φορολογία. Έχουμε στρατηγική μηδενική ανοχής ε, από πλευρά τη Τράπεζα μα για τέτοιου είδους ε, τεχνάσματα φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγής. Δημοσιεύσαμε δε τις εκθέσεις αναχώρα για το 2014 σύμφωνα με τη CDR4 και επίσης η έκθεσή μας για το 2015 ε, θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο. Επίσης, ε, για το 2014 υπολογίζουμε ότι θα συμμορφωθούμε για τις εκθέσεις αναχώρα σύμφωνα με την τυπολογία BEDS δεν προβλέπουμε την προσφορά σύμβουλων για την φοροαποφυγή ούτε σε ιδιώτες πελάτες, ούτε σε επιχειρήσεις, ούτε σε πολυεθνικές. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Το δίνω το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚΑ στην Τανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω και για τους δύο εκπροσώπους των τραπεζών. Θα αρχίσω με την Deutsche Bank. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, στα πλαίσια της φορολόγησης των ε, bonus, των πριμ, έχουμε δει τι γίνεται με τις φορολογικές ε, ρυθμίσεις, αλλά εδώ σκέφτομαι και την περίπτωση ακριβώς αυτών των μπόνους. Η διαφορά ανάμεσα στο νόμιμο και στο ηθικό το νόμιμο που βασίζεται στους νόμους του κράτους και το ηθικό που είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Όταν παρακάμπτει κανείς τον ε, νόμο, μερικές φορές σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οπότε θέλω να ρωτήσω, η δικιά σας σύσταση όσον αφορά τη φορολόγηση των μπόνους, ποια θα ήταν ώστε να είναι πιο σωστό το σύστημα, πιο αποτελεσματικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπο να σχεδιαστεί η νομοθεσία με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε σύγκρουση δύο αυτές αρχές του νόμιμου και του ηθικού δηλαδή. Για την Deutsche Bank είναι η ερώτηση αυτή. Μάλιστα. Δύο λεπτά για να απαντήσετε. Αν κατάλαβα καλά, δύο πράγματα ρωτάτε. Πρώτον, για τις συναλλαγές. Το αναφέραμε ήδη πολλές φορές ότι η... βάσει των δικών μας προδιαγραφών αξιολογούμε τις συναλλαγές που γίνονται βάσει της νομοθεσίας και του κοινωνικού πλαισίου. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στα μπόνους που έχει αναφέρει ο τύπος που πρόκειται για διακανονισμούς όσον αφορά τα μπόνους, πράγματα που γίνανε το 2004. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασε την Deutsche Bank πρόσφατα. Εμείς ε, δεν ε, συμμετέχουμε και δεν στηρίζουμε αυτό του είδους τις ρυθμίσεις στο σημερινό πλαίσιο. Ωραία. Να περάσω τώρα στην Τράπεζα της Σκοτίας. Στα πλαίσια των επενδύσεων που κάνετε, θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από επενδύσεις που γίνονται με φορολογικές απαλλαγές. Αλλά από ό,τι φαίνεται εσείς δεν πληρώσατε τίποτα η μεταρρύθμιση της φορολόγησης της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας, γιατί πρόκειται για ταινίες οποίες ε, επενδύσατε, εσείς τι απαντάτε στην προσέγγιση του ΟΣΑ όπου μπορείτε να επωφεληθείτε εφόσον υπάρχουν δαπάνες από την πλευρά σας στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αποφεύγετε η μέχρι το μέχρι τώρα μοντέλο. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Τι δαπανίσαμε όσον αφορά τις ταινίε και τις συναλλαγές τις οποίες αναφερθήκατε. Το 2006 και το 2007 ήτανε. Επρόκειτο για νόμιμες συναλλαγές με κάποιες φορολογικές αναβολές. Τα συζητήσαμε με τις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και εγκρίθηκαν. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία γενικά, συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία σε ίσχυ και υπάρχει και ο κώδικας διοντολογίας που έχουμε υπογράψει. Οπότε συμμορφωνόμαστε και με το πνεύμα και με το γράμμα του νόμου. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τώρα δουλεύουμε στο ΝΕΣ, το περιβάλλον. Υπάρχουν συναλλαγές που έχουν γίνει παλιά, ιστορικά. Κάποιες που εκείνη την εποχή ήταν νόμιμες συναλλαγές, στα σημερινά πλαίσια δεν θα ήταν πια νόμιμες. Εφόσον δεν τηρούν και το πνεύμα του νόμου και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα έλεγα ότι η σαφήνεια είναι κάτι πολύ βασικό, αλλά καλό είναι να καταλαβαίνει και κανείς γιατί υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Και να την τηρεί αντί να προσπαθεί να την παρακάμψει. Να καταλαβαίνουμε και το θέλει από την νομοθεσία αυτή. Ευχαριστούμε ο Γέπε Κοφούτ που είναι μέλος των σοσιαλιστών και συνεισηγητής. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τις τράπεζες που ήρθαν σήμερα. Θέλω να ρωτήσω και τις δύο τεξής. Πρώτα απ' όλα όλοι έχετε ακούσει για τα Panama Papers που ο τραπεζικός ε, τομέας καθέται στο ειδόλιο και πάλι για σχεδιασμούς επιθετικής φορολόγησης, για φορολογικές ρυθμίσεις και ότι στραβές υπόνοιες γίνονται σε βάρος των τραπεζών σας θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. Μια που είσαστε εδώ λοιπόν θέλω να σας δώσουμε την ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν οι επιχειρήσεις σας έχουν αναμειχθεί καθόλου με την επιχείρηση Μουσάκ Φανσέκα, Φονσέκα που είναι εκείνη τοπική του Παναμά, το δικηγορικό γραφείο ή με κάποια άλλη αντίστοιχη συνεργάζεστε με δικηγορικά γραφεία. Δεύτερον, κάποιος από εσά ξέρει, έχει υπόψη του δικηγορικά γραφεία τα οποία βοηθούν πελάτες των τραπεζών σας και που μπορεί έτσι να βρίσκονται μπλεγμένοι σε αυτή την ε, υπόθεση που αποκαλύπτεται τώρα με τα Panama Papers. Πρόεδρος, ίδια ερώτηση και για τους δύο. Παρακαλώ, εσείς κυρία μου πρώτα. όσον αφορά την ειδική ερώτηση που κάνετε για το δικηγορικό γραφείο του Παναμά. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Νομίζω ότι η υπηρεσία τύπου μας έχει αντιδράσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε ενισχύσει τις διαδικασίες μας όσον αφορά τους πελάτες μας για να μην υπάρχει κανένας ε, μπλεγμένος σε θέματα νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Εμείς δεν βοηθούμε τους πελάτες μας για φοροποφυγή, δεν είναι η πρακτική μας αυτή. Οι πολίτες μας χρησιμοποιούν βέβαια δικηγόρους, ε, οι φοροτεχνικούς που τους βοηθούν για τα φορολογικά τους. Τώρα το άλλο που ρωτήσατε, αν το θυμάμαι καλά, ήταν αν συμβουλεύουμε εμείς τους πελάτες μας για offshore εταιρείε και φορολογικούς παραδείσους. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε ε, offshore banking και στα μέρη εκείνα τα οποία θεωρούνται φορολογική παράδοση, οπότε οι πολίτες μας έχουν σχέση με τέτοιες δικαιοδοσίες, αλλά εμείς δεν τους βοηθούμε σε θέματα ούτε φόρο ούτε τίποτα, γιατί έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές ακριβώς για να μην το κάνουμε ποτέ. Γέπε. Ναι, αλλά για να είμαστε σαφείς για αυτό το θέμα, δηλαδή έχετε σχέσεις με επιχειρήσεις όπως ήταν το Μουσακ Φονσέκα και άλλα τέτοια δικηγοριακά γραφεία στον Παναμά ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Μου το επιβεβαιώνετε αυτό. Είπε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα του Παναμά ή για τους συγκεκριμένους συμβούλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Με ρωτήσατε. Ναι, είπα, με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία ή με άλλη αντίστοιχη που βοηθάει να δημιουργούνται offshore εταιρείε σε φορολογικούς παραδείσους. Όπως είπε και η Deutsche, η έγραψε και η Guardian, δημιουργούνται για νόμιμους σκοπούς. Έχουμε διευκολύνει τους πελάτες μας για να μπορέσουν να φτιάξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ε, μονάδες. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά. Θα αρχίσω για το γενικό ζήτημα της φοροποφυγής και φοροδιαφυγής. Εμείς δεν διευκολύνουμε την ε, φοροδιαφυγή των ε, πελατών μας. Κάποιοι συνεργάζονται στενά με τους ε, συναδέρφους και έχουμε πολλές ενισχυμένες διαδικασίες στη συνεργασία αυτή, ώστε πράγματι να μην διευκολύνουμε την φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το σημείο κίνησης για μας. Τώρα για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας μετά από τη δημοσίευση σχετικών άρθρων, έχουμε τραστή που έχουν σχέσεις με την εταιρεία στην οποία αναφερθήκατε. Η τραστή Business με αυτήν υπήρχαν παλιά τέτοιες δραστηριότητες και στη Γενέβη και στο, στα νησιά Τζέρσι, αλλά υποβάλλεται στις ίδιες αρχές και στους ίδιους κανόνες όπως το γενικότερο πλαίσιο φορολογίας. Οπότε δεν ενθαρρύνουμε την φοροδιαφυγή, ούτε βοηθούμε σε αυτό. φροντίζουμε οι πολιτικές μας να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Έχουμε δύο μονάδες και στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης οι θηγατρικές αυτές που θα φτιάξουμε στο μέλλον θα είναι έτοιμες μέσα στους δύο επόμενους μήνες. Για να καταλάβω. Είπατε ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Τι κάνετε αν έχετε την υπόνοια ότι ένας δικός σας πελάτης ακολουθεί πρακτικές φοροδιαφυγής. Συνεργαζόμαστε με το οικονομικό έγκλημα. Οπότε συνεργαζόμαστε ώστε και οι φορολογικές αρχές και το οικονομικό έγκλημα να ενημερώνονται αν υπάρχουν κάποιες υπόνοιες για τέτοιου είδου δραστηριότητες και με email ενημερώνουμε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία από την Deutsche Bank. Γνωρίζει την έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας που ονομάζεται «Καταχρήσεις φορολογικών παραδείσεων». Δύο τέτοιες έχουν γίνει και λέει ότι 98% όλων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους φοροδιαφεύγουν. Το λέει σαφώς η έκθεσή τους. Οπότε θέλω να μου πείτε εσείς τι νόμιμους ε, λόγους έχουν οι πελάτες σας για να φτιάχνουν σε φορολογικούς παραδείσους τέτοιες offshore εταιρείε. Δεν γνωρίζω αυτές τις ε, αναφορές. Ε, όπως σας είπα, λειτουργούμε σε διάφορους ε, τοποθεσίες για νόμιμους επιχειρηματικούς λόγους και στόχους. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες και επιχειρηματικές δραστηριότητες που γίνονται και για παράδειγμα σε δικαιοδοσίες όπως ε, τα νησιά Καϊμάν ή το τελαγουέρ είναι συχνό φαινόμενο να δημιουργούνται οχήματα τιτλοποίησης ή ταμεία όπου οι επενδυτές θέλουν να συγκεντρώσουν τις ε, επενδύσεις τους ή να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ε, και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν την εμπειρογνωμοσύνη ώστε να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε πελάτες για ε, λόγους δηλαδή εμπορικού δικαίου Ξαναρχόμαστε στον κατάλογο των ομιλητών. Εάν μας μείνει χρόνο θα κάνουμε και κατσιδιάι. ECR, Πύρκο Χόραν Λέναρ. Πύρκο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι στην Deutsche Bank. Το σκέλος ε, των ευρωπαϊκών επενδύσεών σας ε, δράζει στο Λονδίνο και απασχολεί 8.000 ε, υπαλλήλους περίπου και το 2014 να φέρθει απώλεια 2,2 δις ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά δεν δεν ε, κατέβαλε φόρους στην ε, Βρετανία. Την ίδια χρονιά η τράπεζά σας ε, που εδράζει στο Λουξεμβούργο απασχολεί 600 υπαλλήλους και σύμφωνα με εφημερίδες κερδίσατε 49 δις, ε, εκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ στο Λουξεμβούργο. Φαίνεται δηλαδή να είχατε πολύ καλή χρονιά στο Λουξεμβούργο και φρικτή χρονιά στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχω λοιπόν αυτές τις δύο ερωτήσεις για σας. Πρώτον, πόσο φόρο πληρώσατε στο Λουξεμβούργο το 2014. Δύο, πώς ε, ήταν τόσο επικερδής η δραστηριότητα σας στο Λουξεμβούργο ε, σε αντιστοιχεία με πολύ μεγαλύτερες ε, δραστηριότητες και συναλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ θα απαντήσω. Όπως σωστά είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πολύ μεγάλες δραστηριότητες που αφορούν τις παγκόσμιες αγορές, και επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ συν ε, σημαντικές συμβολές από τις άλλες επιχειρήσεις εκτός από την PPC. E στο Λουξεμβούργο ασχολούμαστε περισσότερο με τη διαχείριση πλούτου και περιουσιακών στοιχείων που στηρίζουν τις δανειοδοτικές μας δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο. Η τράπεζα έχει περάσει από δύσκολα χρόνια τα τελευταία διετία και οι απώλειες δεν οφείλονται σε ένα μόνο πράγμα. Ε, σε δύο πράγματα οφείλονται οι απώλειε το 2014 στον ΕΒ. Το ένα είναι γενικά η κατάσταση τη αγορά, της παγκόσμια αγορά, και έπειτα ε, λόγω των κανόνων για την αποκάλυψη των στοιχείων στις εκθέσεις ένα χώρα δείχνουμε εισοδήματα από συναλλαγές ανάμεσα στους ομίλους που δεν, διασυνοριακά που δεν διαγράφονται στις ε, δηλώσεις των ομίλων. Το Λουξεμβούργο είχε καλά λειτουργικά αποτελέσματα και πιο σταθερά αποτελέσματα από το 2014. Δεν επηρεάστηκε από τις αναταραχές των αγορών στις επενδυτικές αγορές και τις παγκόσμιες αγορές. Όσον αφορά τους φόρους που καταβάλαμε, στο Λουξεμβούργο ανέρχεται στο 28% για το 2014 και νομίζω έτσι απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Φάβιο Ντεμάζη από την ΚΟΕ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στη Deutsche Bank. Την ερώτησή μου. Επιβεβαιώνεται ότι επηρεάζεστε από την Panama Leaks και οι μη γερμανικές σας επιχειρήσεις είναι ακριβώς η κόμβη που λειτουργούν πάνω-πάνω ε, 10 ε, της λίστας. Είστε στο Λουξεμβούργο εσείς. Ε. Πριν από λίγες εβδομάδες ρώτησα για τον Παναμά, εγώ και μου είπαν μα δεν ξέρω τίποτα για τον Παναμά γιατί δεν έχω ιδέα. Τώρα μου είπατε ότι πρέπει να διαβουλευτείτε με τους πελάτες σας πρώτα. Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί χάνουμε χρόνο και νομίζω ότι παίρνετε αρκετά καλό μισθό για να έρχεστε εδώ και να παριστάνετε ότι δεν ξέρετε τίποτα και δεν έχετε να μας πείτε τίποτα. Είστε σε θέση να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις, ε, τις ερωτήσεις των συναδέλφων που δεν απαντήσετε. Ε, αυτή είναι η πρώτη μου απλή ερώτηση. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω πόσα χρήματα έχετε βάλει στην άκρη για τις νόμιμες διαδικασίες που σχεδιάζονται με τη φοραποφυγή, τη νομική συμβουλή, δηλαδή, εφόσον όλα αυτά τα κάνετε για επιχειρηματικούς σκοπούς και διερωτώ με, ε, άμα βλέπουμε τα έγγραφα του Παναμά, τι σημαίνει επιχειρηματικούς σκοπούς, να φτιάχνετε ε, εταιρείε ε, για αυτούς που ασχολούνται με την παιδική πορνεία. Αυτό είναι business για σας. Τι θα πει business purpose, επιχειρηματικό σκοπός. Τέλο, tax ruling στο Λουξεμβούργο 2009 και 2010. Μπορείτε να μας πείτε πόσες ακόμα, πόσα ακόμα ειδικέ φορολογικές ε, ρυθμίσει έχετε λάβει από τότε μέχρι σήμερα. Επίσης, από τα 800 εκατομμύρια φτάσατε σχεδόν σε 1,6 δις ευρώ ε, στο Λουξεμβούργο. Πώς έγινε αυτό και πόσες, πόσες είναι οι εταιρείε που εσείς ρυθμίσατε να στήσει η Μονσέκ για λογαριασμό των πελατών σας. Uh, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν μπορώ να δώσω εγώ ε, στοιχεία για νόμιμα αποθεματικά. Ναι, αλλά ε, εάν δεν ασχολείστε με την ε, φορολογική, εάν δεν κάνετε φοροδιαφυγή, τότε θα ήταν μηδενικά αυτά τα αποθέματα. Μου είπατε για ξέπλυμα χρήματος και νομικά ζητήματα. Δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένες υποθέσεις. Τότε γιατί είστε εδώ, ρωτάει κάποιο. Τι θα μας πείτε. Υπήρξαν τέσσερις ειδικέ φορολογικές ρυθμίσεις σε σχέση με το LuxLeaks Αυτό που ζητάμε είναι φορολογική βεβαιότητα για θέματα όπου οι νόμοι περί φορολογίας δεν εξασφαλίζουν αυτή τη βεβαιότητα και τα ακούσαμε και σήμερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να βασιστούμε. να ξέρουμε τι είναι τα rulings, αυτές οι ειδικέ ε, φορολογικές αποφάσεις. Αλλά πόσες ε, είχατε από το 2010 και μετά. Δεν νομίζω πως είναι σχετικό. Πρόεδρος, Ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι βουλευτής εκλεγμένος. Εγώ αποφασίζω αν είναι, έχουν σχέση οι ερωτήσεις μου ή όχι. Πρόεδρος, η κυρία έχετε το λόγο. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών στο Λουξεμβούργο, έχουμε αυξημένα επιχειρησιακά αποτελέσματα στο Λουξεμβούργο του 2015 Επίσης βλέπετε ότι το ποσοστό φορολόγησης ήταν χαμηλότερο στο Λουξεμβούργο το 2014 και 2015 και αυτό λόγω του κύκλου εργασιών μας και του EBIT, το που είχαμε και δραστηριότητες που υπόκειται σε μηδενική φορολόγηση. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε γραπτά απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεν απαντήσατε και πότε. Εγώ απάντησα νομίζω πλήρως ερωτήσεις. Όχι, όχι, δεν απαντήσατε πλήρω, λέει ο Πρόεδρο. Εγώ θέλω να επανέλθω σε δύο από τι ερωτήσει. σω να υπήρξε μια παρεξήγηση. Για τα rulings ο κύριος Δετομάση θέλει να ξέρει πώς ε, υπήρξαν. Εσείς λέτε ότι όχι, δεν είναι σημαντικό το νούμερο αυτών. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί τότε, εάν το λέτε αυτό. Και θα πρέπει να εξηγήσετε κιόλα και αυτό ενδιαφέρει το συνάδελφο, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα rulings που έγιναν κάποτε και τα πιο πρόσφατα. Αυτό είναι το νόημα της ερώτησης. Μπορείτε να απαντήσετε. Δεν έχω τις πληροφορίες, θα σας απαντήσω γραπτά. Μια εβδομάδα προδιορία για να απαντήσετε γραπτός. Δίνω τώρα το λόγο στην Μόλι Σκοτ κάτω από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, εμένα η ερώτησή μου απευθύνεται στην ε, Τράπεζα της Σκοτίας. Από μια απτική βρετανική, αν θέλαμε να δούμε ποιε είναι οι φορολογίες ε, για τους πλούσιους και τους πολλά έχοντες στη Βρετανία, θα στραφούμε προς την UBS και την ΚΑΤΣ ε, στην Βρετανία. Αυτό που δείχνουν τα έγγραφα του Παναμά ε, ε, είναι ότι η πλειοψηφία φτιάχτηκαν, οι εταιρείε μάλλον, οι πλούσιοι μάλλον, στα νησιά της ε, Μάγης. Δηλαδή η ίδια, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να φτιάξει offshore ε, εταιρείε και βλέπουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην καρδιά αυτής της ε, βιομηχανίας ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Η ΚΟΤΣ επίσης ε, έχει, ζητήσει, έχει στήσει 500 εταιρείες offshore στο Τζέρσι και μάλιστα ήταν η έβδομη πιο δημοφιλής τράπεζα που χρησιμοποιούσε αυτές τις υπηρεσίες για να θεσπίσει εταιρείε, για να στήσει μάλλον εταιρείε. Επειδή εσείς είστε εκπρόσωπος της Τράπεζας Σκοτίας, θα θέλαμε να μας πείτε σε ποιο βαθμό η τράπεζά σας ήταν αναμειγμένη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, που οδήγησε σήμερα σε αυτό το σκάνδαλο. Κούτς, Ηνωμένο Βασίλειο, Κούτς, ε, Τζέρσι και UPS, Τράπεζα της Σκοτίας, ε, Βρετανία και Τζέρσι. Πώς όλα αυτά συνδυάζονται με την απόφασή σας να γίνετε απλή, απλούστερη, ισχυρότερη και πιο δίκαιη. Επίσης, πώς η τράπεζά σας στηρίζει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο Τζέρσι όταν διχειρίζετε τα χρήματα πλουσίων ανθρώπων. Πώς γίνεται. Μήπως επειδή ακριβώς σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους είναι πιο εύκολο να κρύβετε το τι κάνετε. Τώρα, επειδή η τράπεζά σας θα είχε πτωχεύσει το 2008 αν δεν είχε ρίξει ένα σωρό χρήματα το κράτος και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτήτη το κράτος κατά 73%. Πώς εσείς προσφέρετε τέτοιου είδους υπηρεσίες στους πλούσιους στους να τη στιγμή που έχουμε τεράστιο πρόβλημα και το έλλειμμά μας διαρκώς ε, αυξάνεται. Ε, ε, υποβαθμίζεται το σύστημα υγείας, κλείνουν βιβλιοθήκες. Εσείς βοηθάτε τον πλούσιο κόσμο να ξεφεύγει από την φορολογία. Πώς γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σας ευχαριστώ. Να σας πω λίγα πράγματα πρώτα για το τι κάνουμε στο Τζέρζι; Έχουμε μια υπεράκτια τράπεζα που λέγεται RBS International που κατ' ουσίαν είναι μια πλήρης ε, τράπεζα επενδυτική και λιανική. Οι βασικές της δραστηριότητες είναι απλές τραπεζικές υπηρεσίες δανεισμού, καταθέσεων, πληρωμών και η RBSI επίσης ε, διευκολύνει τραπεζικές υπηρεσίες για άτομα τα οποία κινούνται διεθνώς. Αυτό ακριβώς ε, βρίσκεται στο Τζέρσι. Αυτό είναι κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει. Όσον αφορά την ΚΟΥΤΣ, οι διεθνείς της δραστηριότητες που όπως σωστά είπατε κατέληξαν σε μια ρύθμιση σύμφωνα με το, τον Συμβασμό Ελβετίας και ΕΙΠΑ έλαβα ε, μια στρατηγική απόφαση να πωλήσουμε την Κούτς και όσον αφορά τις μελλοντικέ μας λειτουργίες ε, θα διατηρήσουμε μια λειτουργία ιδιωτικής ε, τραπεζικής ε, την Κούτς, δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όπως είπα υπάρχει και η Κούτς ε, στο Τζέρζι. Και όπως σας είπα παίζει και ρόλο θεματοφύλακα. Όπως είπα και πριν, η λειτουργία του θεματοφύλακα συμμορφώνεται με τους κανόνες που υπάρχουν ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, όπως και όλη η τράπεζά μας. αυτό είναι τμήμα της ε, φιλοσοφίας μας και για το μέλλον. Όσον αφορά το περίπλοκο της κατασκευής, Εδωμέν της ιστορίας της τράπεζας, προφανώς ε, είχαμε μια σειρά εξαγορών ε, άλλων τραπεζών και τώρα απλοποιούμε. Αλλά η RBSI, η RBS International δηλαδή, δεδομένου του ότι παρέχει πλήρης υπηρεσίες του Τζέζι που ρυθμίζεται πάρα πολύ θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας Γνωρίζουμε βεβαίως ε, το τι πρέπει να κάνουμε και προσπαθούμε πάντα να συμμορφωνόμαστε με τις αρχές ε, και πολιτικές που ήδη ανέφερα όσον αφορά την φοροδιαφυγή και την διευκόλυνση της ε, φοροαποφύγης. Σας ευχαριστώ για το διευθυντή ο Μαρκοτσάνη. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω την ερώτησή μου προς την κυρία της Deutsche Bank. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτό το οποίο ακούσαμε πριν το, την απαράδεκτη ερώτηση. Απαράδεκτο είναι το ότι έχετε πλήρη πρόσβαση για να κάνετε lobbying, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έρχεστε εδώ πέρα και αρνείστε να απαντήσετε στους συναδέλφους. Εάν, όπως λέτε, θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα ήθελα τουλάχιστον να απαντάτε στις ε, ερωτήσεις μας. Ε, δεν έχουμε την απέτηση να τις ξέρετε όλες τώρα τις απαντήσεις, μπορείτε όμως να απαντήσετε γραπτός. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις ε, μεταξύ του σελβετικής ε, ε, θηγατρικής σας και της εταιρείας Asset Management Mosset στις Αντίλες κατόπιν. Τι γίνεται με τα Profit Participating Instruments. Ποια οικονομική λογική έχουν αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η Deutsche Bank και θα ήθελα επίσης να αντιληφθώ τον ρόλο των συμβούλων για μεγάλες εταιρικούς πελάτες. είναι δηλαδή το συγκεκριμένο συμφέρον της ε, Deutsche Bank για να συμμετέχει σε τις μα Και η τελευταία ερώτηση αφορά την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας. Οι εκθέσεις αναχώρα δείχνουν μεγάλες ε, διαφορές ε, ανάλογα με την χώρα στην οποία δουλεύει ο κάθε υπάλληλο. Π.χ. στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους αποδίδουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Πώς έχετε και τόσο μεγάλες ε, διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ Γερμανίας και Ιρλανδίας ή Γερμανίας ε, και νήσων ε, Καϊμανή άλλων τέτοιων χώρων. Σας ευχαριστώ. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Μπορείτε λίγο να διευκρινίσετε την ερώτησή σας για την ελβετική θηγατρική. Ναι. Για τα Panama Leaks μιλάω βλέπουμε εκεί πέρα πως ε, η ελβετική θηγατρική σας ε, είχε σχέσεις ε, με την εταιρεία Mosfon SA η οποία είναι θηγατρική της Mosfon Fonseca. Μπορείτε λοιπόν να διευκρινίσετε την σχέση μεταξύ της ελβετικής ε, θηγατρικής ε, και της εταιρεία ε, Mosek Fonseca. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να απαντήσω και ζητώ συγγνώμη αν δεν τα καταφέρνω. Δυστυχώς δεν γνωρίζω ε, για τι γίνεται με την ελβετική θηγατρική. Ναι, ναι, ευχαριστώ. θα σας απαντήσω γραπτός. Όσον αφορά τα profit participation instruments, Πρόκειται για κάποια αξιόγραφα τα οποία σύμφωνα με την αίσθηση στο παρελθόν μετρούσαν ως ε, ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1. Νομίζω πως με τους νέους κανόνες θα καταργηθούν, ναι, θα θεωρούνται πλέον tier 1. Δεν παρέχουν κάποιο ιδιαίτερο φορολογικό πλεονέκτημα. Υπάρχει μια συμμετρία μεταχείρισης της ε, τράπεζας και του επενδυτή. Όσον αφορά τις ε, εκθέσεις αναχώρα, θεωρούμε πως οι εκθέσεις αυτές, όπως φαίνεται και στη έτη 2014 και 2015, δίνουν μια καλή εικόνα της ε, λειτουργίας μας, της 70 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Όσον αφορά την παραγωγικότητα, πρέπει να αντιληφθείτε πως έχουμε διαφορετική σύνθεση σε κάθε χώρα. Στην Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη, παρέχουμε υπηρεσίες υποδομών και παγκόσμιες τραπεζικής που οπωσδήποτε έχουν άλλο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τη διαχείριση πλούτου ή το private banking στη Γερμανία οπωσδήποτε ακολουθούμε τις ε, διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές ε, για το transfer pricing του ΩΣΑ. Αυτό νομίζω φαίνεται. γιατί τα κέρδη μας φαίνονται στις χώρες στις οποίες υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Και οι εκθέσεις αυτές, αν δείτε την κερδοφορία μόνο ένα αριθμό υπαλλήλων δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη. Εγώ λοιπόν θεωρώ πως ακολουθούμε αυτές τις διεθνείς ε, κατευθύνες γραμμές και το ίδιο ισχύει και για την κερδοφορία που παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστώ. Τα, τα ακουστικά σας βγάλετε λίγο. Για το τελευταίο ερώτημα του κ. Τζανί είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε με πολλές τράπεζες. Και πρέπει να δούμε ότι σε αυτή τη νέα απάντηση και απέτηση για τις καταχώρα εκθέσεις, τελικά οι τράπεζες είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί ο νόμος τις υποχρέωσε πριν από οποιαδήποτε άλλη πολυεθνική οντότητα να κάνουν την δημοσίευση αυτή και να είναι και διαθέσιμη για το κοινό. Ένα από τα πράγματα που μας εξέπληξε είναι ότι σε ορισμένες τράπεζες, αν κάνουμε έναν υπολογισμό παραγωγικότητα, τζίρος, ανά υπάλληλο, υπάρχει τεράστια διαφορά χώρα. Οπότε θα σας συμβούλευα τις τράπεζες γενικά και μεθαύριο και τις άλλες πολυεθνικές που θα κληθούν να κάνουν το ίδιο, να το λάβετε υπόψη σας στην ετήσια έκθεση. Γιατί όσο πιο συχνά υπάρχουν ε, κανονικές επεξηγήσεις που συνάδουν με τη φυσιολογική λειτουργία μιας τράπεζας, μιας πολυεθνικής, εντάξει, αλλά μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που να είναι πιο επίμαχοι. Το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με όλες τις τράπεζες και συμπληρώνω βασικά την απάντησή σας. Ίσως λοιπόν στις ετήσιες εκθέσεις σας θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Τώρα, ο κύριος Μπερνάρ Μονό έχει το λόγο από την Ευρώπη των Εθνών και τη Ελευθερίας προς την ε, Ερμπές. Αγοράσατε την τράπεζα Σκούτς και για ένα διάστημα ακολουθήσατε τις ελβετικές πρακτικές. 40 δις ήταν το ποσό το 2008, κάτι το οποίο πλήρωσε και Ευρωπαίος φορολογούμενος. Κάθε φορά που εσείς ή μια άλλη τράπεζα καταδικάζετε για φορολογικές απάτες, πάντα απαντάτε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή λέτε τι πρακτικές έχετε εφαρμόσει, τι καλές είναι τώρα και ότι ποτέ δεν θα ξαναγίνει το ίδιο. Όμως ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, οι πρακτικές αυτές. Χτες είχαμε νέο σκάνδαλο, Panama Leaks. Ε, μην μπω σε λεπτομέρειες, προφανώς δεν θα φταίτε, γιατί έκτοτε έχετε ενισχύσει τις ε, διαδικασίες σας. Όμως, οι τράπεζες κάθε τόσο στριμώχνονται ποτέ οι διευθύνσεις σας δεν προλαβαίνουν τα πράγματα και δεν φροντίζουν εκ των προτέρων να έχουν κάποιες τεχνικές για να αποφύγουν τέτοιου είδους σκάνδαλα. Οπότε ρωτάω, η στρατηγική σας τετολογία περιλαμβάνει και τον κίνδυνο αμαύρωσης της εικόνας σας. Και η τράπεζά σας δεν φοβάται ότι τελικά οι πελάτες θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εσά, όπως επίσης και οι διάφορες χώρες. Ο Διευθυντής για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την φήμη, τον κίνδυνο, την έλλειψη εμπιστοσύνη. Τα γνωρίζουμε, η τράπεζά μας τα ξέρει και έχουμε πολύ ψηλές προδιαγραφές. Και η Διοκτησία φροντίζει να υπάρχει συμμόρφωση. Έχουμε πολύ δυνατούς ελέγχους για να αποφεύγουμε και την φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους. Εντάξει, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάτι να πάει στραβά. Η στρατηγική μας όμως και η επιθυμία μας είναι να είμαστε μια πιο απλή και σωστή τράπεζα και να απομακρυνθούμε από κάθε στοιχείο που έχουμε κληρονομήσει που θα παραβίαζε τους σημερινούς κανόνες. Η διεύθυνση είναι σαφής πάνω σε αυτό. Και όταν πρόκειται για την φοροδιαφυγή, για μας κάτι τέτοιο είναι εντελώς απαράδεκτο. Το ίδιο και όσον αφορά την φοροαποφυγή και των τραπεζών δεν διευκολύνουμε ούτε τους ε, πελάτες μας, ούτε στις συναλλαγές μας έχουμε τέτοιες πρακτικές. Δεν αποτελεί μέρος της ηθικής της τραπεζάς μας. Θέλουμε φυσικά να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών μας στην τραπεζά μας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε με τους ελέγχους και τις πολιτικές που έχουμε εγκαθιδρύσει στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστούμε. Η Ντανούτα Χιμπνερ, εκ μέρους του ΑΛΚ. Θέλω να ρωτήσω και τις δύο τράπεζες να απαντήσουν στην ερώτησή μου, παρακαλώ. Πολλές συναντήσεις είχαμε ήδη με συναδέλφους σας από άλλες τράπεζες και κάθε φορά που δίνουμε παραδείγματα ερευνών που γίνονται όσον αφορά τη φοροποφυγή την φοροδιαφυγή, ακούμε ότι πρόκειται για το βάρος του παρελθόντος για πράγματα που έχουν κληρονομήσει τράπεζες από το παρελθόν. Και εσείς είπατε το ίδιο και είπατε ότι τώρα μπαίνετε σε μια νέα περίοδο ε, συμμόρφωσης με τους κανόνες και μέτρων να που Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα τέτοιων μέτρων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και σε εθνικό επίπεδο. Οπότε θέλω να ξέρω εσείς οι τράπεζές σας τι μπορούν να κάνουν ώστε να διασφαλίσουν ότι τέτοιες περιπτώσεις φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής δεν θα επαναλαφθούν και ότι αυτό το βάρος του παρελθόντος δεν θα εξακολουθεί να επηρεάζει το μέλλον. Τι μέτρα φαντάζεστε ότι μπορούν να ληφθούν κώδικας δοντολογίας ή κάτι άλλο. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων μέτρων. Πρώτε κυρίες, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως είπα και εισαγωγικά, εμείς έχουμε κώδικα δεντολογίας και ηθικής εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Τις αρχές αυτές και τις αξίες και τα πιστεύω τα έχουμε συμπεριλάβει στην αξιολόγησή μας όσον αφορά τις συναλλαγές μας και έτσι ξέρουμε τι παραμέτρους επιτρέπουμε στις συναλλαγές δεν είναι τόσο ότι έχουν αλλάξει οι εσωτερικές μας ε, διαδικασίες, γιατί πάντα φροντίζαμε για την ε, χρηστή διαχείριση. Περισσότερο έχει να κάνει με αξίες και πιστεύω στο κοινωνικό επίπεδο. Πώς δηλαδή βλέπει κανείς τις συναλλαγές. Μιλήσαμε πολύ για το νομικό. Εννοείται ότι οι συναλλαγές πρέπει να είναι νόμιμες ό,τι συναλλαγές έχουμε είναι νόμιμες. Σήμερα κοιτάμε και τα πιστεύω μας και τις αξίες μας τεχνικά. Δηλαδή κοιτάμε να δούμε και τι είναι σωστό, τι είναι καλό. Και λαμβάνουμε και αυτό υπόψη για να αξιολογήσουμε μία συναλλαγή μας. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Ωραία, προσλήψεις, αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω. Έχετε διαφορετική προσέγγιση τώρα για τις προσλήψεις πώς ε, επιλέγετε το προσωπικό σας ώστε να είσαστε σίγουροι ότι θα τηρήσουν τις αρχές αυτές. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, για είναι θέμα του τομέα προσλήψεων αυτό, ότι αν οι υπάλληλοι μας δεν τηρούν τις αρχές και τα πιστεύω αυτά, παίρνουμε αυστηρά μέτρα. Και δρούμε ανάλογα. Με όλους τους υπαλλήλους φροντίζουμε οι αρχές και τα πιστεύω αυτά να εφαρμόζονται και διασφαλίζουμε ότι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι εννοούμε με αυτά. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ. Για μας αρχίζουμε με την πρακτική αξιολόγηση των τραπεζών προκειμένου να συμμορφώνονται προς τον νόμο οι ίδιοι έτσι λαβαίνουμε υπόψη μας διάφορες αρχές. Και θέλουμε οι αρχές αυτές να ισχύουν στις συναλλαγές. Και όλες οι πλευρές, όλες οι τράπεζες, όλοι, όλες οι διακλαδώσεις των τραπεζών να τηρούν τις αρχές αυτές. Είτε πρόκειται για νέα προϊόντα, είτε για νέα, νέου είδους συναλλαγές, να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι αρχές. Στη συνέχεια εντοπίζουμε τους φορολογικούς σχεδιασμούς και έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με προειδοποίησεις σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένους τραπεζίτες που κλιμακώνουν κάπως την κατάσταση. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις και ελέγχουμε να δούμε κατά πόσο η συναλλαγή έγινε βάσει των αρχών μας ή όχι. Αν είναι αποδεκτή ή όχι. Κοιτάμε επίσης και τις Επιτροπές Νέων Προϊόντων που τους ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Να ρωτιόμαστε το ίδιο πράγμα κατά πόσο οι πρακτικές που ακολουθούν είναι αποδεκτές. Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, ήδη είπα ότι είναι στοιχείο κλειδί το φορολογικό τμήμα και το, και το οικονομικό έγκλημα συνεργάζονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν ε, υπόνοιες που έχουν εκφραστεί. Όσον αφορά τις προσλήψεις, θα έλεγα ότι έχουμε κάποιες αξίες κλειδί, οι οποίες αποτελούν μέρος της λειτουργίας μας. Τις έχουμε υιοθετήσει και αποδεχτεί. Και κάθε φορά που έρχεται κάποιος να δουλέψει σε εμά, φροντίζουμε να είναι αποδεκτές και γι' αυτόν οι αρχές αυτές. Νίνα Γκίλ, λοιπόν, εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα την RBS και την απάντηση που μόλις δώσατε. Σαν κούφια λόγια μου ακούγονται γιατί είδα την σελίδα σας και λέτε ότι ε, έχετε στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των φορολογικών ζητημάτων και την συμμόρφωση με το φορολογικό δικαίωμα αλλά με βάση τα όσα ακούσαμε χτες με τα Panama Papers πραγματικά θεωρώ ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι πολλοί από τους πελάτες της Mosset Fonseca συναλλάσσονται μαζί σας ε, και είχαν εταιρείε που ήταν ε, σε, αυτές, σε αυτές τις χώρες. Και πολλές αρδανικές τράπεζες έχουν τέτοιες θηγατρικές και οι RBS. Πέρσι είχαμε μια έκθεση που έδειχνε ότι η RBS έχει 404 θηγατρικές σε φορολογικούς ε, παραδείσους. Δηλαδή δεν συμβάζονται αυτά τα πράγματα και μόλις μας είπε μια συνάδελφος ότι πληρώστε 23 εκατομμύρια ευρώ στο γερμανικό κράτος για να συμβιβαστείτε για μια έρευνα φοροδιαφυγής ναι, την Κούτς και πραγματικά αυτό το οποίο μου τη δίνει είναι ότι ένα στέλεχος ε, ηχογραφήθηκε να λέει ότι κοιτάξτε οι φορολογικές αρχές είναι ο εχθρός και ε, μιλάμε για μια τράπεζα η οποία ακόμα είναι στην ιδιοκτησία του κράτους, κατά 73%. Πώς δικαιολογείται λοιπόν το να εργάζεστε σε φορολογικούς παραδείσους όταν πολλοί φορολογούμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους λόγω το, της λιτότητας και των περικοπών στα επιδόματα και τις υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα πληρώνεται 5 εκατομμύρια μπόνους στην διοίκησή σας και άλλα 70 εκατομμύρια σε μελλοντικά μπόνους. Ενώ ταυτόχρονα έχετε ζημία 2 δισεκατομμύρια το 2015. Θεωρείτε λοιπόν πως οι τράπεζες θα πρέπει ε, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες φορολογικού συστήματος για να αποκτήσουν κάποιο πλέον έκτημα. Γιατί λέτε, επίσης πολλοί λένε ότι εμείς δεν δίνουμε τις συμβουλές, αυτό το κάνουν οι τέσσερις μεγάλες ε, ελεγκτικές εταιρείε. Ποια είναι η σχέση σας με αυτές και πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Και τελευταία μου ερώτηση. Θα δεσμευτείτε για περισσότερη διαφάνεια για να μην μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα από διαρροές. Και ποια είναι η ε, θέση της ε, τράπεζάς σας για να δίνει λογαριασμό στο κοινό αναχώρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ερώτηση για την RBS. Να ξεκινήσω από την ερώτηση για τους φορολογικούς παραδείσους. Όπως είπα, μειώνουμε τον αριθμό των θηγατρικών μας και αυτό θα περιλαμβάνει και αρκετές ε, χώρες με χαμηλή φορολογία και στο τέλος της υπόθεσης αυτής θα έχουμε θυγατρικές μόνο σε χώρες και περιοχές ε, οι οποίες εξαρτώνται από το βρετανικό στέμα που υπάρχει επαρκής ρύθμιση. Τα υπόλοιπα σχόλια δεν μπορώ να πω ε, κάτι. Δεν ε, θεωρώ πως η ερώτηση αυτή ήταν εντός του πλαισίου της Επιτροπής όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Για το θέμα της εκμετάλλευσης ε, των αδυναμιών στην νομοθεσία, οπωσδήποτε όχι. Εμείς ακολουθούμε το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Δεν προβάλλουμε σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είτε για εμάς είτε για τους πελάτες μας. Για τις μεγάλες τέσσερις εταιρείε ε, τις λογιστικές, ναι, ε, τις χρησιμοποιούμε. για πράγματα τα οποία δεν, μπορεί να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εσωτερικά. Ο προπολογισμό μας για υπηρεσίε ε, συμβουλών το 2014 ήταν 8 εκατομμύρια λίρες ε, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια πήγαν σε ζητήματα που αφορούσαν την διευθέτηση με το προσωπικό και τα υπόλοιπα 5 αφορούσαν την αναδιάρθρωση της τράπεζας για την διαφάνεια. Έχω ξεκαθαρίσει πως ε, είμαστε οπωσδήποτε δεσμευμένοι για την ασφάλεια για τις εκθέσεις αναχώρα δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα του 2014 αναχώρα και το ίδιο θα γίνει και στην έκθεση βιωσιμότητας του 2015. Και βέβαια το BEPS ε θα το υφθήσουμε το 2016 και μετά. Κύριε Διευθυντρία. Μπορείτε να τα επαναλάβετε. Ναι, ναι. θεωρείτε πως οι τράπεζες θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα σημεία του φορολογικού συστήματος ε, για ε, τους δικούς τους σκοπούς ε, και ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αν θα, κάνετε, θα υποβάλλετε εκθέσεις χώρα; Η απάντησή μου νομίζω θα συμφωνήσει με του συναδελφού. Χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες συμβούλων εκεί όπου δεν έχουμε την δική μας ε, πείρα ή δεν εκπροσωπόμαστε, δεν έχουμε δικό μας φορολογικό τμήμα. Για τις εκθέσεις αναχώρα και διαφάνεια είμαι υπέρ. Έχουμε πλήρη διαφάνεια απέναντι στις φορολογικές αρχές και ευχαρίστω συμμορφωνόμαστε όσον αφορά την διαφάνεια και συμμορφωνόμαστε οπωσδήποτε και με όλους τους νόμους και τις απαιτήσει ε, διαφάνειας και ιδιαίτερα βεβαίω ε, όσον αφορά την BEPS ε, και τις ενισχυμένες εκθέσεις αναχώρα. Για την πολιτική μας και τις διαδικασίες μας, όπως είπα, Θεωρώ πως ο κόσμος έχει αλλάξει και θεωρώ πως οι συναλλαγές μας γίνονται εντός των φορολογικών μας αρχών και του κώδικα ηθικής έτσι ώστε να είναι σύνομες αλλά να θεωρούνται ε, και ηθικές θα έλεγα και για να προστατεύσουμε όλες και την φήμη της εταιρεία μας. Σας ευχαριστώ. Πέρφανος Πέρες. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου απευθύνεται στην Deutsche Bank. Με εντυπωσίασε πολύ στι 5 Σεπτεμβρίου του 2007, πριν από πολλά χρόνια δηλαδή, όταν ο γενικός διοικητής, ο ε, τη Άκερμαν της Deutsche Bank πρώτος είχε πει ότι οι τράπεζες έπρεπε οπωσδήποτε να επιβάλλουν διαφάνεια όσον αφορά την έκθεσή τους στο κίνδυνο. Πιστεύετε πως αυτή η νοοτροπία έχει διεισδύσει σε ολόκληρη την εταιρεία και αν ναι, πώς. Διαπιστώνω ότι το περασμένο Νοέμβριο οι Financial Times αποκάλυψαν ε, ένα τέχνασμα σύμφωνα με το οποίο η Deutsche Bank παρενέβαινε από την Αυστρία και η Βραζιλία για να φτιάξει ένα μηχανισμό Profit Participating Instrument αντίθετο προς τις συστάσεις του ΩΣΑ και του G20 επί το οποίο η Deutsche Bank είχε αρνηθεί να εξηγηθεί, να δώσει εξηγήσεις, μπορείτε σήμερα να μας δώσετε εξηγήσεις. Είπατε ότι για τις εκθέσεις αναχώρα δεν έχετε πρόβλημα. Όντως, Υπάρχουν ε, νομοθεσίες που σας, υποχρεώνουν, υποχρεώνουν να το πράξετε, όμως ε, μπορεί να λειτουργείτε στη Μάλτα πολύ μικρό προσωπικό, λίγο προσωπικό ή στο Γκένζε χωρίς καθόλου προσωπικό. Σε έναν από τους προηγούμενους ε, ερωτώντες είπατε ότι εκεί είναι πιο προσοδοφόρες από ότι άλλες αυτές οι δραστηριότητε. Όμως το φορολογικό ζήτημα εκεί δεν έχει να κάνει για την απόφαση ε, για το πού θα τοποθετηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Ε, τρίτη ερώτηση. Για τα rulings δεν θελήσατε να μας δώσετε λεπτομέρειες. Μας δώσετε πολύ γενικόλογες απαντήσεις, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ακριβώς αν υπήρξαν ε, τέτοιου είδους αποφάσεις ε, ruling ε, με την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Τελευταία μου ερώτηση. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε ότι 17,9% των κερδών σας γεννώνται σε μέρη που μπορούμε να ορίσουμε ως φορολογικούς παράδεισους. Αυτό δεν εξηγεί καθόλου την κατανομή αυτών των δραστηριοτήτων. Δηλαδή δεν το λαμβάνετε αυτό υπόψη. Και, και πάλι, τι αιτιολογεί το ότι 17,9% των δραστηριοτήτων σας ή των κερδών σας γεννάτε σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Η κυρία φορολογικους παραδεισους ευχαριστω κυρια Μπούμου. Να σας απαντήσω για την ερώτηση για τη Βραζιλία πρώτα. Είναι κάτι στο οποίο, το οποίο αναφέρθηκε για το πολύ καλό παράδειγμα για το ε, πώς έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές. Υπήρξαν κάποιες συναλλαγές που συζητήθηκαν με τους πελάτες ή τις επιχειρήσεις αρχικές συζητήσεις. Ωστόσο, στη, καθώς αυτά τα προϊόντα και οι συναλλαγές περνούσαν από τη διαδικασία έγκρισης, πέρασαν από τα διάφορα τμήματα, όπως γίνεται με όλα μας τα νέα προϊόντα, τα απορρίψαμε και τελικά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδου ε, δραστηριότητε στη Βραζιλία και στην Αυστρία. Τότε, ναι, νομίζω πως οι Financial Times σωστά το ανέφεραν ότι ε, απερίφθησαν στο τέλος αυτές οι συναλλαγές. Δεν εγκρίθηκαν και δεν έγιναν ποτέ στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρων, να πω δύο λόγια για τη Μάλτα, γιατί ήταν επίσης ε, πολύ προφανές στη μελέτη που έγινε για τις εκθέσεις αναχώρα το 2014. Ιστορικά, Έχουμε μία τραποζική μονάδα στη Μάλτα. Έχουμε επίσης χρηματοδοτικές δραστηριότητε για τους πελάτες, αλλά και δραστηριότητε εσωτερικής χρηματοδότησης. Επίσης έχουμε ξένες θηγατρικές στη Μάλτα, για τις οποίες, από τις οποίες λαμβάνουμε ε, μερίσματα. Πριν από τρία χρόνια αποφασίστηκε ότι οι δραστηριότητε της Μάλτας δεν ήταν πια στις βασικές μας δραστηριότητες, οπότε αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε από τη Μάλτα και σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες για το, μέχρι το 2020 θα έχουμε κλείσει πια τις επιχειρήσεις μας ε, στην Μάλτα. Όπως σας είπα, κυρίως πρόκειται για ε, μερίσματα από θηγατρικές και από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Μάλτα που δεν χρειάζεται πολύ FTE επιτόπου. Στο Γκένζι έχουμε ακόμα ε, επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Νομίζω πως έχουμε στο Γκένζι FTE, έχουμε δραστήριες ε, επιχειρήσεις βασικά σχετίζονται με τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες για ενδιάμεσες, ε, ομίλου. σύμφωνα με την έκθεση του 2015 το 17,9% αυτό ανεφέρθη στις εκθέσεις 2014, ε, δηλαδή η Deutsche Bank υποτίθεται κινδυνεύει, ε, μάλλον σε μεγάλο βαθμό μεταφέρει τα κέρδη στις ε, δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης. Αλλά τα πορίσματα της έκθεσης δεν είναι σωστά γιατί συμμορφωνόμαστε με τις διεθνείς αρχές, με τιμών μεταφοράς. Το 2014, αν δείτε το συνολικό μας ε, φορολογικό φόρτο, ανήλθε στο 46% που είναι πολύ σημαντικό και αν δείτε τις ε, δηλώσεις ε, τις φορολογικές, αν δείτε το συνδυασμένο ποσοστό, με βάση τη γεωγραφική θέση των κερδών, ο φόρος αυτός είναι 34%, δηλαδή πολύ πάνω από την κρατική φορολογία της Γερμανίας που είναι 31%. Δεν μετακινούμε δηλαδή κέρδη τεχνητά σε, σε, σε ε, δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης μόνο και μόνο για λόγους φοροαποφυγής. Η Deutsche Bank δεν ανέφερε 1,8 δις κερδών σωστά εντός της Ένωσης όμως η έκθεση δεν έδωσε ενημέρωση όσον αφορά το σημαντικό κομμάτι αυτών των εσόδων που θα έπρεπε να πάει σε φόρους και σε δικαιοδοσίες υψηλής φορολογίας όπως τις είπα, που ανέρχεται η φορολογία στο 40%. Και πάλι τέτοιου είδους ισχυρισμοί δεν μπορεί να αποδεικνύουν την υπόθεση αυτή ότι τεχνητά μετακινούμε το κέρδη μας προς δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης. Είχατε τα ruling με το Λουξεμβούργο. Ναι, βεβαίως έχουμε. Και άλλες δικαιοδοσίες στην Ευρωζώνη. Est-ce que, au titre Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των τραπεζών εάν θεωρούν ότι τα καταπιστεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης ε, για να χρησιμοποιηθούν για φοροδιαφυγή και να καλύψουν και άλλες ε, εγκληματικές δραστηριότητες γιατί θεωρείτε ότι η Βρετανική κυβέρνηση αντιστάθηκε. Δεν ήταν η μόνη. Ήταν αυτή η οποία αντιστάθηκε περισσότερο στην συμπερίληψη των καταπιστευμάτων στην ε, οδηγία για την καταπολέμηση του ξεφλήματος χρήματος. Για την αποκάλυψη του, ε, των πραγματικών διοκτητών. Ναι, κοιτάξτε για την χρήση καταπιστευμάτων μπορώ να πω ότι ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους ε, νομιμότατους ε, σκοπούς μεταξύ των οποίων διαχείριση και προστασία διαφόρων στοιχείων η κληρονομιά και έτσι χρησιμοποιούνται και για εμάς για να διαχειριστούμε ακριβώ τον κίνδυνο ε, και αν υπάρχει όπως είπαμε κάποια χρήση η οποία δεν είναι σωστή επανερχόμαστε στους κινδύνους ε, που ε, υπάγονται στο καθεστώς του ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον πελάτη μας και το τι θέλει να κάνει. Πράγματι μπορούν να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους. Τώρα δεν μπορώ. Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη. Για το θέμα αυτό. Και για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να θέσει ερώτηση στους ε, προσκεκλημένους μας. Ναι, Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα μαθαίναμε περισσότερα αν είχε γίνει συνεδρία σε αυτή και, κλεισμένων των θυρών. Θέλω να ξέρω γιατί δεχτήκατε αυτήν την συνάντηση, γιατί ήρθατε, ενώ στο τέλος τώρα έχουμε την αίσθηση ότι αρνηθήκατε να μας δώσετε νέες πληροφορίες σε σχέση με όσα ήδη ξέρουμε από τον τύπο, από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς τι θέλετε να κρατήσουμε εμείς σαν νέο στοιχείο που μας φέρατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Ο Διευθυντής πρώτα και μετά κυρία. Συγγνώμη, δεν άκουσα την αρχή της ερώτησης. Επαναλαμβάνει η κυρία Μπερές. Θα λέγατε περισσότερα αν ήμασταν και κλεισμένο το θυρών. Όχι, είναι η απάντηση. Θα απαντούσαμε τα ίδια, ακριβώς τα ίδια. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας όσο καλύτερα μπορούσα. Όχι, δεν θα έκανα διαφορά. Δεν θα Ήταν διαφορετικές οι απαντήσεις μου. Τώρα όσον αφορά το τι προσφέραμε στη σημερινή συζήτηση, θα έλεγα τους τρόπους με τους οποίους βοηθάμε τις διεθνείς επιχειρήσεις να συμμορφώνονται καλύτερα στους κανόνες. Από εκεί και πέρα, αν σε κάτι δεν ήμουν ασαφής, ευχαρίστως, ρωτήστε με να σας απαντήσω. Σίγουρα εμεί δεν βοηθάμε τους πελάτες, όπως είπαμε, να προβαίνουν σε αθέμητες πρακτικές φορολογικές. Αυτό είναι το βασικό. Εσείς, για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις συναντήσεις Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Είναι καλό να υπάρχει διάλογος μεταξύ μας για το πώς έχουν αλλάξει οι πρακτικές μας, οι φορολογικές μας αρχές. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας απέναντι στις φορολογικές αρχές και απέναντι του κοινού. Ελπίζω να το, αντιληφθήκατε αυτό, κυρίως μετά το Panama League... Εγώ έχω λίγε πληροφορίες στα χέρια μου βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά ευχαρίστω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Επειδή μόλις έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε αυτό το θέμα, δεν έχω ακόμα αρκετέ πληροφορίες στα χέρια μου. Και από εκεί πέρα, αν είμαστε και κλεισμένα των θυρών, και εγώ το ίδιο έχω να πω ότι δεν θα είχα απαντήσει διαφορετικά στι ερωτήσει σα. Προεδρό. ωραία, ο εισηγητή μα θα καταλήξει σε συμπεράσματα. Τι σχόλια θα μπορούσαμε να πούμε στους προσκεκλημένους μας. Αυτά που σας ρωτήσαμε είναι μερικά από αυτά που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Και θα σας τεθούν από εδώ και πέρα και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πελάτες σας, από τους μετόχους σας και από τους ίδιους τους φορολογούμενους και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ακούσετε πολλές ερωτήσεις ακόμα. Κυρίως όσον αφορά τις αποκαλύψεις τώρα από τα έγγραφα αυτά του Παναμά. Θα διευκρινιστούν τα πράγματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε, καλά θα κάνετε να είσαστε όσο γίνεται πιο ξεκάθαροι, απλοί στις απαντήσεις σας, να απαντάτε με διαφάνεια. Ε, προφανώς εδώ οι ευρωβουλευτές δεν ικανοποιήθηκαν απόλυτα. Τώρα επιπλέον από αυτά που μας είπατε, υπενθυμίζω κυρίως για την Deutsche Bank ότι μας χρωστάτε μια γραπτή απάντηση στην ερώτηση του κύριου Ντεμάζη που δεν είναι εδώ για τη διαφορά στις φορολογικές ρυθμίσεις πριν και μετά. Πριν και τώρα ουσιαστικά. Είπατε ότι αυτό που ήταν ε, σημαντικό δεν ήταν τόσο αριθμός όσο το περιεχόμενο. Οπότε πολύ θέλουμε να ξέρουμε αυτό το περιεχόμενο, πώς άλλαξε η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν, για παράδειγμα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Επίσης μας είπατε ότι θα μας απαντήσετε γραπτά και για τις σχέσεις της Ελβετικής Θηγατρικής και τις σχέσεις της με την Μοσέκ Φονσέκα του Παναμά. Είπατε πίσω ότι δεν μπορούσατε να απαντήσετε, αλλά το καταλαβαίνουμε φυσικά απόλυτα, για κάτι που σας ρώτησε η κυρία Εύα Ζόλη, για πριν από χρόνια βέβαια, όσον αφορά τις επικρίσεις στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια ακρόασης που έγινε εκεί. Η κυρία Βαζολή έκανε μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Αν θέλετε γραπτά να σας πει πιο συγκεκριμένα τι εννοούσε. Παρακαλώ. Νομίζω πως ε, δεν αφορούσε γενικά μια ακρόαση με την Deutsche Bank. Ήταν μια γενικότερη ακρόαση. Κοιτάξτε, προτείνω να το διευκρινίσει γραπτός. Βεβαίω. Κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τις δύο τράπεζες που ήρθαν σήμερα εδώ για την συζήτηση αυτή. Για μένα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα η ίδια η δουλειά της τράπεζας. Είστε μεγάλες ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τώρα έχετε τις εκθέσεις αναχώρα και ελπίζουμε αυτό να γίνει παγκόσμια υποχρέωση για όλες τις εταιρείες αλλά δεύτερο και σημαντικό σε σχέση με τα Panama Papers είναι το πως οι τράπεζες χρηματοπιστωτικός κλάδος γενικότερα, η, τα δικηγορικά γραφεία κλπ. να βοηθούν άτομα, πολυεθνικές επιχειρήσεις να αποφύγουν φόρους ή να φοροδιαφύγουν. αυτό το οποίο είδαμε με τα Panama Papers είναι μία εταιρεία μόλις, η Μουσάκ Fonseca. Mm. Ναι, αλλά ξέρουμε πως υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες. πρέπει λοιπόν και εσείς να τηρήσετε αυτό το οποίο είπατε περί ηθικής. Πρέπει αυτό το οποίο είπατε λοιπόν να το τηρήσετε κιόλας. Και στην έκθεση την πρώτη της Επιτροπής μας είχαμε κάποια ξεκάθαρα συμπεράσματα για τις λογιστικές εταιρείες, για τις τράπεζες, κατευθυντήρες γραμμές, για το πώς ε, μπορούν οι εταιρείε αυτές να δραστηριοποιούνται, αλλά νομίζω πως ε, και χρειάζονται και επαρκείς κυρώσεις. Αν δηλαδή οι τράπεζες ή άλλες εταιρείες εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες, αποφυγής και φοροδιαφυγής ε, θα μπορούσαν οι κυρώσεις να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Π.χ. πρόστιμα ή να μην συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακραίες περιπτώσεις να αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας. Υπάρχει συγκεκριμένο, συγκεκριμένη νομοθεσία. Ελπίζω λοιπόν ζητήστε κι εσείς δημοσίως ε, κάποια νομοθεσία για να υπάρχουν σοβαρές ε, συνέπειες στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Σιγητέ, Ευχαριστώ άλλη μια φορά τους ε, προσκεκλημένου. Ολοκληρώσαμε την εξέταση ημερησία μας διάταξης. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 18 Απριλίου για αυτή τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση 3 με 6.30. Πέρα συνεδρίαση.